Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μια πρόταση, επειδή μόλις ήρθε ο κύριος Τζαμπάσκι, έχουμε 13 λεπτά τελικά, ένα τέταρτο, για να εξετάσουμε την έκθεσή του. Θα έλεγα λοιπόν να το δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο. Κύριε Τζαμπάσκι, έχετε το λόγο. Уважаеми και κύριοι, θα ήθελα να σας ε, θυμίσω ότι το 2007 υπήρχε ένας κανονισμός ο οποίος εγκρίθηκε ο 697 του 2016 είχε να κάνει με την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία τους από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο κανονισμός τώρα αυτός, ο GDPR, θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018. Υπάρχει ο κανονισμός 45 του 2001 και ο 679 του 2016. Οι, οι δύο κανονισμοί αυτοί ε, πρέπει να ευθυγραμμιστούν και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν σταλεί οι αναγκαίες αλλαγές για την έγκριση του κανονισμού του 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μας παρουσίασε ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη δουλειά τους. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένες ε, τροπολογίες, πολύ συγκεκριμένες, πολύ ευαίσθητες. Αφορούν την μετάδοση δεδομένων και η παρούσα πρόταση αποκλίνει από τον κανονισμό. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, συγκατάθεση, ε, την ε, την, τους ανηλίκους και το όριο Ε, νομίζω πως μετά την ψηφοφορία του Σεπτεμβρίου θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε στην Επιτροπή μία πολύ καλή δουλειά, ένα επικοδομητικό κείμενο το οποίο θα προστατεύει τα ε, δικαιώματα των πολιτών για τα προσωπικά τους δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, πολύ καλά. Ο κύριος Άξελ Βός έχει στήσει το λόγο, παρακαλώ. Θα προσπαθήσω... και εγώ να είμαι σύντομος. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση και για τους προβληματισμούς τους οποίους ε, παρουσιάζετε. Θα ήθελα να σταθώ ίσως σε δύο-τρία σημεία. Ε, για εμάς ε, το ΕΛΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό η, η εξέταση της αναλογικότητας υπό το άρθρο 9 ε, παράγραφος 1β να διατηρηθεί και να μην αντικατασταθεί από διάφορα άλλα συμφέροντα. Να τηρηθεί η αναλογικότητα λοιπόν. Για μας αυτό είναι μία από τις προτεραιότητές μας και αν επιθυμείτε θα μπορούσαμε και εμείς να προτείνουμε μία διατύπωση. Μετά, αυτό που θεωρούμε αρκετό, αρκετά σημαντικό έχει να κάνει με τα δεδομένα για διοικητικού σκοπού, τα διοικητικά δεδομένα και τα επιχειρησιακά δεδομένα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ε, αρμόδιες για ποινικά ζητήματα, Europol, Eurojust. Εκεί θεωρώ πως είναι σημαντικό να γίνει μια διάκριση Τώρα το ύψος ε, των ε, προστήμων, εάν θα πρέπει να επιβάλλονται ή όχι, ε, αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν νομίζω πως είναι ίσως καλό ένα θεσμικό όργανο να επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα σε κάποιο άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε όλα αυτά έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλες τις ε, λεπτομέρειες, να, είναι, να είμαστε πολύ ακριβείς σε σχέση με τους ορισμούς και ιδιαίτερα ε, με, τον ορισμό, ε, με τον κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς. κυρία Ρέκνερ, όχι. Ο κύριος, κυρία Μπερζεγό, ούτε. Μάλιστα. Κύριε Τζαμπάσκη, έχετε το λόγο. Α, ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέλει να πει κάτι. Είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια μεταξύ τη πρόταση ε, μεταξύ του κανονισμού για τα θεσμικά όργανα τη Ένωση και του γενικού κανονισμού. Ε, προσπαθήσαμε λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα δύο όργανα, ε, τα δύο κείμενα. Το μόνο σημείο που μπορεί να υπάρξει μια απόκληση είναι η αυξημένη προστασία ε, για τους πολίτες με βάση την εμπειρία που είχαμε από την εφαρμογή του υπάρχους κανονισμού του 47 2001 εδώ και 15 χρόνια. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τις, ε, τα πρόστιμα είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας, είναι θέμα αρχής. Όπως σε εθνικό επίπεδο μπορεί να επιβληθούν λοιπόν πρόστιμα στους δημόσιους φορείς, έτσι λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δείξει το καλό παράδειγμα. Ε, θα πρέπει δηλαδή και αυτή να μπορεί να τους επιβάλλονται πρόστιμα. Αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριο Τζαμπάσκη παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους ε, και σας κύριε Φως για τα σχόλια. Θα τα αναλύσουμε και θα επανέλθουμε. Πολύ ωραία. Κλείσαμε και με το σημείο αυτό. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά, πέντε λεπτά με την ψηφοφορία. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να είναι και όλοι εδώ. Και επειδή έχουμε πει ότι θα ψηφίσουμε στις 10, θα περιμένουμε. Chers collègues, mesdames, messieurs, comme euh, nous l'avons annoncé. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Έδωσα χρόνο στους συναδέλφους να πάρουν θέση. Σας θυμίζω ότι η ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Φεράρα αναβλήθηκε για την 28η στην Επιτροπή Γιούρη και θα ξεκινήσουμε τώρα με την ψηφοφορία, την πρώτη ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Ρέγκνερ. Παρακαλώ να έχετε ετοιμάσει τις κάρτες σας και να είστε έτοιμοι εφόσον χρειαστεί. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται ένα ζήτημα με τη διερμηνία προς τα αγγλικά. Α, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Έκθεση λοιπόν της κυρίας Ρέγνερ, τροπολογία 32. Είστε έτοιμοι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Μετρήσατε, τα καταφέρατε. Ξαναρχίζουμε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Επειδή είναι τεράστια η αίθουσα... Ε, υπέρ. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ θα πάει πιο γρήγορα ηλεκτρονικά μάλλον κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Α, συγγνώμη, 7, 35 και 36 από κοινού. Μάλλον 7 και 35 πρώτα. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Πέρας ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Δεν ξέρω αν η κυρία, η κυρία ψήφισε. Ναι, πολύ ωραία. Ε, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Όχι, συγγνώμη, ναι, ήταν εντό των, της προηγούμενης ψηφοφορίας. 34. Α, όχι. Συμβαστική 1. Άρχισε ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λείπει μια ψήφος. Πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 39. Άρχιτη ψηφοφορία. Μας λείπει ακόμα κάποιος. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Προφορική τροπολογία. Θέλει κάποιος το λόγο. Όχι. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Αν λείπουν δύο. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Παρακαλώ, ναι. Ναι, με όλο το σεβασμό δεν υπάρχει υποχρέωση ψηφοφορίας. Ε, και όταν ε, γίνεται έτσι και περιμένουμε τελευταία στιγμή, κάνουμε τρεις φορές περισσότερο χρόνο να ψηφίσουμε. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά χρειάζεται να είμαστε και ευγενείς. Αν δεν έχετε κάποιο τρένο και δεν βιάζεστε, καλό είναι να περιμένουν να ψηφίζουν όλοι. Αν έχετε αντίρρηση, πράγμα. Εγώ θα ακολουθήσω τη γραμμή σας, βέβαια, αν είστε κάθετα αντίθετοι. Λοιπόν, μου λένε ότι αν ένας βουλευτής δεν θέλει να συμμετάσχει στην ψηφοφορία, απλά αφαιρεί την κάρτα του. Και έτσι δεν χρειάζεται να ε, περιμένουμε. Ωραία. Σαράντα τρία. Όχι, συγγνώμη, 42, δεν ψήσαμε τροπολογία 42. Α, καταπίπτει μάλιστα. 43, 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Άρχεται ψηφοφορία. ψηφίσετε όλοι. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 3. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη, καταπίπτει. Τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται. Συμβιβασμό 4. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπο... Ε, Συμβασμό 5, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρα ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε ονομαστικά επί του συνόλου άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Ρέγνερ. Και τώρα θα περάσουμε στην δεύτερη έκθεση. Πάλι της κυρίας Ρέγνερ. Είστε έτοιμοι. Τροπολογία 42. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 43. Άρχεται. Ψήφισαν άπαντες πέρα Απορρίπτεται. 9. Και 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες πέρα. 10 και 46. 47 μάλλον. 10, 46 και 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν το... Πέρας. Ε... Τώρα περνάμε στη συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 50. Άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 14. Άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. 53 άκτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 και 54. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 και 55. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 και 56. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 και 7 ε, άρχεται, πέρας, εγκρίνεται. 20 21 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 άρχεται. Απορρίπτεται. 23 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 25 και 25 και 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 59. Ε, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 60. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 1. Πρώτη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2. Άρχεται. Πέρας. Αγκρίνεται. 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Καταπίπτη. Έχετε δίκιο. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 4. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 4.35. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 7 και τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 41. Άρχεται η ψηφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Le vote est clos. Ah. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στην κυρία Ρέγνερ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Χρυσογόνου. Ιστολέτιμη, τροπολογία 35. Ο κύριος Μπούντα για προφορική τροπολογία ζητά το λόγο. Ο κύριος Φώστα θα μιλήσει εκ μέρους του. Εκπροσωπώ λοιπόν τον ε, κύριο Μπούντα, ο οποίος έχει υποβάλει μια προφορική τροπολογία για την τροπολογία 23. Εκεί αναφέρεται η λέξη sentencing, η οποία αντικαθίσταται με τη λέξη conviction. Sentencing δηλαδή, αυτή η λέξη πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη conviction. Pas d'opposition. Nous passons au vote. Euh. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αντιρρήσει. Περνάμε στην ε, ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία. 35. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίβεται. 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 42. Άρχεται η ψηφορία. να άπαντε. Πέρας. Απορρίπτεται. 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 47. Άρχεται την ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 50, ε, άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 51. Άρχισε η ψηφοφορία. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι. 51. Ε, άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πενήντα Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 55. Νομίζω εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Διότι στην τροπολογία 55 λέει ότι καταπίπτει εάν εγκριθεί 55. Κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον την 56 εννοεί, τέλος πάντων κάτι τέτοιο. Η 56 εάν ε, εγκριθεί πίπτη. Αντώνιο έχεις δίκιο. Όπως απορρίφθηκε, ψηφίζουμε ό,τι και αν γίνει την 55. 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. 57 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 58 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα του 61. Άρχεται η ψηφοφορία. 61 δεύτερο τμήμα και 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 62. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 63. Άρχεται. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται επίσης. 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Εξής ανάπαντες πέρας. Απορρίπτεται. 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται 74 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 75 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 76 άρχεται η ψηφοφορία Εψήφισαν άπαντες πέρας. Απορρίπτεται. 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνεται. 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Απορρίπτεται. 79 άρχεται. Πέρας. Εγώ δόντα. Ε, υπέρ. Μέλλον άρχεται, πέρας, απορρίπτεται. 81 άρχεται, πέρας, εγκρίνεται. 82 82 άρχεται. Εψήφισαν παντέ εγκρίνεται. 83 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ένα, Συμβαστική ένα, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 15. Προφορική τροπολογία. Κύριε Μπούντα. Μάλλον κύριε Φως. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Φως. Είναι μια προφορική τροπολογία στην 15, ε, όπου 15 θέλουμε να προστεθεί εξή διατύπωση στο τέλος του κειμένου που θα λέει αυτό θα δημιουργούσε ενισχυμένο νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία αποτελεσματικότερα και να περιοριστεί η απειλή από τρομοκρατικές οργανώσεις ώστε να γίνει δυσκολότερο για αυτές να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση για την προφορική τροπολογία του κυρίου Μπούντα. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Κάνω μια μικρή οπισθοδρόμηση με την αδειά σα. Μου είπαν ότι δεν ψηφίσαμε την 83 που είναι ακριβώ από πάνω. Ψηφίστηκε η 83. Συμφωνούμε και απορρίφθηκε. Οπότε λύθηκε το θέμα. Συνεχίζω με τη 15. Πάμε στη 16. Άρχεται. Πέρα. Αγκρίνεται. 17. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 18. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 19. Άρχεται. Συμβατή με την 18 έτσι καλλιώς. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 19. Άρχεται. Ναι, αλλά μου ζητήθηκε χωριστή ψηφοφορία. Αφού είναι συμβατή με τη 18, φαντάζομαι θα ψηφίσετε το ίδιο. Οπότε άρχεται η ψηφοφορία. Για να μην υπάρξουν μετά αντιρρήσει. 19 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. 20. Άρχεται. Να να άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 22. Άρχεται. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. 23 με προφορική τροπολογία του κυρίου Μπούντα που θα μας πει ο κύριος Φως. Όρος sentencing να αντικατασταθεί από το conviction. Πολύ ωραία. Περνάμε στην ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 προφορική τροπολογία. Φαντάζομαι με τον ίδιο τρόπο κύριε η προφορική τροπολογία για την 25. όπου υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στους νομικούς ορισμούς για τα υποκειμενικά στοιχεία που απαιτούνται για να καταρτιστεί ε, δίκημα. Αλλά αυτοί οι ορισμοί δεν έχουν ε, θεωρηθεί επαρκές ουσιαστικό πρόβλημα για την διασυνοριακή συνεργασία. Έτσι θα διαμορφώσει το κείμενο η προφορική τροπολογία. Εμείς προτιμάμε το πρωτότυπο, χωρίς την προφορική. Να ψηφίσουμε για την απόρριψη της τροπολογίας της προφορικής ή μια και καλή. Εγώ θα έλεγα να ψηφίσουμε για την τροπολογία. Οπότε ψηφίζουμε για την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ πολύ. 26. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εκρίνεται. 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 29 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Τροπολογία πρώτη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται δύο άρχεται πέρας εγκρίνεται τρία άρχεται πέρας Απορρίπτεται. 4. Πέρας. Απορρίπτεται. 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 7 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 32 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 33 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Άρχεται. Πέρας. Και τελικ... απορρίφθηκε και τώρα τελική ψηφοφορία ε, ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Ρέγνερ. Φοβήθηκα για λίγο. Ναι, συγχαίρω την κυρία Ρέγνερ, ενώ πρέπει να συγχαρώ, τον κύριο Χρυσόγωνο. συγγνώμη. Η κυρία Ρέγνερ εδώ κοκκίνησε από την τροπή της και σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πάλι συγγνώμη. Και τώρα περνάμε στο σημείο 13 για την νομική βάση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία. Πρώτη τελευταία. Συγγνώμη. Για την αναδιατύπωση. Εγώ είμαι εισηγητής. Όχι, ο κύριο Μαστάλκα είναι τελικά. Υπάρχει εδώ μια αντιστροφή. Να ψηφίσουμε το κύριο Μαστάλκα πρώτα. Α, και τα δύο είναι ο κ. Μαστάλκα, μάλιστα. Πρώτα το σημείο 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα, ψηφίζουμε εκ νέου, δεν υπήρξε πρόβλημα με την ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα επί του 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Μαστάλκα. Σας ευχαριστούμε για την ηλεκτρονική αυτή ψηφοφορία. Ήταν πιο απλό για να μπορούμε να είμαστε ακριβείς. Ένα μικρό διάλειμμα λίγα δευτερόλεπτα και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης. Merci. <laughs> Έχουμε καθυστερήσει, συνάδελφοι, οπότε περνάμε στο σημείο 16. Θα ήθελα όμως πριν ε, να αναφερθώ στο που είπε η κυρία Ρέντα, η οποία θέλει νομίζω να ε, κυματογραφήσουμε την συζήτηση, την παρέμβασή της, δεν έχω τη λάβει ακριβώς. Ναι, αν δεν έχετε αντίρρηση, υπάρχει εδώ ένα μέλος των Πρασίνων που θα βιντεοσκοπήσει την παρέμβασή μου, αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Έχει κανείς αντίρρηση? Έχετε πολλούς φίλους, βλέπω, κανείς δεν αντιτίθεται. Πολύ ωραία. Όχι, σοβαρά Έχει κάποιο αντιρρήσει. Ο κύριος Βόλκιν έχει το λόγο. Για τις 330 τροπολογίες. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε 330 περίπου 323 τροπολογίες και αυτό δείχνει πόσο διαφορετικές απόψεις έχουμε για το μέλλον της ψηφιακής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ όμως ε, πάρα πολύ για αυτές τις τροπολογίες. Ε, οι διατάξεις του άρθρου 2 είναι από τις πιο επίμαχες. Πολλές τροπολογίες ζητούν διαγραφή του άρθρου ε, μέχρι και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Ιδιαίτερα Υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί από αρκετούς συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες, από κοινού λοιπόν για ε, να επανεξετάσουμε την ε, αρχή. Ε, μετά από τις επιτροπές ΙΤΡΕ, Ίμκο και Κούλτ υπάρχουν ε, πολλές διαφορετικές απόψεις και συμβιβαστικές προτάσεις έτσι ώστε να βρούμε μία λύση. Θα ήθελα λοιπόν ε, να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία για να σας ε, παρουσιάσω τις δικές μου κόκκινες γραμμές για τον κανονισμό. Η απλουστευμένη πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα μέσω διαδικτύου είναι ένα κεντρικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς είναι ένα θέμα το οποίο ε, έχει συμφωνία από όλες τις ε, πολιτικές απόψεις και έχει να κάνει για την ποιότητα της ε, δημοσιογραφίας. Η ποιότητα της δημοσιογραφίας είναι πάρα πολύ σημαντική για την διασφάλιση της αντικειμενικότητας. Οι συνάδελφοι κυρίως από το ΕΛΚ επιχειρηματολογούν υπέρ της οδηγίας για την πνευματική ιδιοκτησία λέγοντας ότι χρειάζεται ενίσχυση της προστασίας ιδιαίτερα απέναντι στο πρόσφατο φαινόμενο των fake news. Υπάρχουν σχετικές τροπολογίες οι οποίες ε, αφορούν το θέμα αυτό ε, για ε, τους, για τους οργανισμούς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς, ιδιωτικούς οι οποίοι πρέπει να ε, προστατευτούν. Δεν χρειάζεται λοιπόν αποδυνάμωση των κανόνων, το αντίθετο ενίσχυση. Χρειάζεται όμως γι' αυτό μία χωρίς ε, σύνορα καθολική πρόσβαση στη, στο τηλεοπτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Υπάρχει επίσης μια κατανόηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει συμφωνία ότι θέλουμε να προχωρήσουμε την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς. Ε, η ελευθερία του τύπου δεν πρέπει σε, και η ελευθερία της άποψης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζονται. Γι' αυτό χρειάζεται γρήγορη ε, και ε, αξιόπιστη πρόσβαση στο περιεχόμενο, ακόμα και αν κάποιος βρίσκεται σε διαφορετική χώρα. Ε, γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης να πω ότι ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι, κυρίως νέοι, ε, απολαμβάνουν το ρετιλοπτικό περιεχόμενο μέσω διαδικτύου και όχι μέσω των τυπικών επιγραμμικών μεθόδων. Γι' αυτό χρειάζεται και μία προσαρμογή της ε, δικής μας στάσης. Υπάρχει λοιπόν και είναι πολύ γνωστό αυτό ε, σε όλους και στην βιομηχανία μια πολύ μεγάλη ε, ανάγκη για να αλλάξουν τα πράγματα και επίσης σε ό,τι αφορά ε, τις αμοιβέ, τις διατάξεις περί αμοιβών, τις ρήτρε που αφορούν την το forum shopping, την αναζήτηση της πιο ευνοϊκής δικαιοδοσίας, πρέπει να τις κοιτάξουμε. Θεωρώ πως η ψηφιακή εσωτερική ε, αγορά έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και ε, πρέπει όμως αυτό να γίνει με σεβασμό στα ε, δικαιώματα των πολιτών και με βελτίωση της πρόσβασή τους στο ε, το τηλεοπτικό περιεχόμενο, ιδιαίτερα για εκείνους που ζουν σε μεθοριακές ε, περιοχές. Η Επίτροπος Βεστάγκερ μαζί με τους ε, σκιώδες ηγητές και εμένα έχει συζητήσει πολλές φορές, ιδιαίτερα μάλιστα την περίπτωση Sky. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να συμμετέχουν όσοι το επιθυμούσαν. Κρατήσαμε έναν πάρα πολύ κλειστό κύκλο. Όσοι όμως επιθυμούν μπορούν να ενημερωθούν γιατί ε, είμαστε στη διάθεσή τους. Το μήνυμα που αποκομίσαμε από όλες τις ε, συζητήσεις είναι ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στον κανονισμό και την υπόθεση Sky. Έχει ζητηθεί όμως να περιμένουμε το τέλος της ε, υπόθεσης έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο νομοθετικό μας έργο. Και σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Υπάρχουν επίσης και κάποια ερωτήματα που προκύπτουν. Ε, καταρχάς, όλες σχεδόν οι πολιτικές ομάδες ζήτησαν τα τεχνικά ε, προβλήματα που αφορούν την ε, απευθείας διαβίβαση να ρυθμιστούν. Επίσης υπάρχουν πολλές φωνές που ζητούν το θέμα αυτό να χειριστεί σε εθνικό επίπεδο. Μετά, ε, κάτι που αφορά κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ρήτρα για εφάπαξ ε, αμοιβή θα ισχύει και για ραδιόφωνο μετά. Ε, αυτά προς το παρόν. Να ευχαριστήσω ξανά τους και εισηγητές και όλους τους συναδέλφους για τις ε, τροπολογίες που υπέβαλα. Νομίζω πως αυτό θα κάνει τη δουλειά μας ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει το λόγο. Κυρία Βρέντα. Ρέντα, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καθα... καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή προεπεξεργασία του κειμένου, του σχεδίου έκθεσης. Αυτό το θέμα είναι επίκαιρο. Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα μόλις έλαβα πάρα πολλές επιστολές και υπογραφές από πολίτες που... Ε, μου είπαν ότι ναι, ήθελα και εγώ να δω την ε, διαμάχη για τις ε, γερμανικές εκλογές μεταξύ των δύο κύριων υποψήφιων, αλλά δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα γιατί βρισκόμουν στη λάθος πλευρά των ε, συνόρων. Και πολύ περίεργα δεν μπορούσαν να το δουν σε κάποιες σε κάποιες περιπτώσεις στο διαδίκτυο ακριβώς λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων στη Γερμανία. Αυτό δείχνει πως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά καθόλου τα προβλήματα της κινηματογραφικής ε, βιομηχανίας μόνο. Αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, είναι διασυνοριακό και άκρος πολιτικό. Χρειαζόμαστε όλη η πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε πολιτικά θέματα. Οι Γάλλοι μάλιστα ε, μας έδειξαν ότι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ε, δική μας ε, προεκλογική ε, περίοδο και αυτό ε, καταρχάς είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε πως κάποιος άλλος λαός ενδιαφέρεται για την ιστορία μας και είναι ε, παράδεκτο να υπάρχουν εμπόδια και φραγμοί μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη. Πρέπει να υπερπηδήσουμε αυτά τα εμπόδια και α μην ξεχνούμε κιόλα πω υπάρχουν και γλωσσικέ μειονότητε. Για παράδειγμα, η γερμανική γλωσσική μειονότητα στη Δανία και στο Βέλγιο, οι οποίοι δεν έχουν τώρα τη ε, δυνατότητα να δουν ε, προγράμματα στη γλώσσα του, ε, ακόμα και αν το επιθυμούν. Και μάλιστα μόνο σε τρεις-τέσσερις ε, χώρες υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε video on demand. Ε, γερμανικών προγραμμάτων. Δεν υπάρχει λοιπόν καν η δυνατότητα να έχει κάποιος πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα και δεν τίθεται θέμα ε, εσόδων φυσικά. Δεν μπορείς να έχεις έσοδα εάν δεν δει κάποιος τη δουλειά σου. Μετά, οι γλώσσες είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Βλέποντας ε, ξενόγλωσσα προγράμματα μαθαίνεις γλώσσα. Ε, στην περίπτωση μου υπάρχουν πάρα πολλοί που μαθαίνουν γερμανικά βλέποντας τηλεόραση. Να μην ξεχνάμε επίσης και τους καλλιτέχνες οι οποίοι ε, χάνουν ε, απολαβές από πνευματικά δικαιώματα επειδή ακριβώς δεν μπορεί να προβληθεί το περιεχόμενό τους ε, πέρα από τα σύνορα της χώρας τους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης από το διαδίκτυο σε αυτά τα προγράμματα, ιδιαίτερα κυρίως μάλιστα από την δημόσια τηλεόραση και να δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή στους ε, νέου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, δεν υπάρχουν αρκετά προγράμματα για εκείνου και πόσο μάλλον διαθέσιμα και στο διαδίκτυο. Ε, τώρα, συμφωνώ απόλυτα με ε, την άποψη του εισηγητή για το ότι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι ουδέτερη είναι, και πρέπει να είναι απόλυτα επιγραμμική. Όταν δηλαδή κάποιος έχει τη δυνατότητα επίγεια να ε, βλέπει τηλεόραση, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το κάνει και αυτό από το διαδίκτυο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απευθείας διαβίβαση, θα ήθελα να πω ότι έχουμε υποβάλει σχετικές ε, τροπολογίες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως εμείς πιστεύουμε πως χρειάζεται ρύθμιση εδώ, αλλά χρειάζεται συγκεκριμένες προτάσεις για τα προβληματικά σημεία χωρίς να χρειαστεί να ορίσουμε εκ νέου τα πράγματα. Υπάρχει, όπως, είπε και, υπάρχει, όπως ακούσαμε και η αντίστοιχη οδηγία τα πνευματικά δικαιώματα, τις οποίες εισηγητής είναι ο φως και εκεί θα δείτε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Και είναι άκρος προβληματικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν δύο ε, προτάσεις, δύο νομοθετήματα, τα οποία θα λένε διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε υποβάλει ε, και εγώ προσωπικά τροπολογίες, τις οποίες θα βρείτε ε, και από την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ε, αφορούν λοιπόν αυτήν την απευθείας ε, διαβίβαση και θα ήθελα στο τέλος να αναφερθώ στην άγρα δικαιοδοσία ε, και τις απολαβές. Εγώ θεωρώ πως οι απολαβές θα πρέπει να είναι ανάλογες της, του έργου που προσφέρουν Χρειάζεται όμως εδώ προσοχή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ε, ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών οι οποίοι ε, θα χρησιμοποιούν προγράμματα τα οποία έχουν άδεια για παράδει... και θα τα ξαναπέζουν για παράδειγμα στις ε, ειδήσει. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια προσοχή στη ρύθμιση σχετικά με τις απολαβές των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων. Και σε ό,τι αφορά αυτό το forum shopping, νομίζω πως αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει υπάρχει στο χαρτί, δεν υπάρχει ουσιαστικά. Οι οργανισμοί ραδιοτηλεόρασης δεν μπορούν να αλλάξουν για παράδειγμα την έδρα τους για να πάνε σε μια διαφορετική χώρα ε, και έτσι να ξεπεράσουν τα προβλήματα του γεωγραφικού αποκλεισμού. Η διατύπωση τώρα του εισηγητή σε ορισμένα σημεία είναι κάπως επικίνδυνη, διότι με τη διατύπωση που χρησιμοποιεί μπορούμε, ε, μπορεί να επηρεαστούν ε, τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι εκπέμπουν σε παραπάνω από μία χώρα. Για παράδειγμα, ο σταθμό Άρτε που εκπέμπει και στη Γαλλία και στη Γερμανία με δίγλωσο πρόγραμμα. Ε, αυτά από μένα. Να ευχαριστήσω ξανά θερμότατα τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε και να πω πως ελπίζω να ολοκληρώσουμε ε, αυτήν την έκθεση σύντομα έτσι ώστε να αποφεληθούν όλοι οι χρήστες στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας, ο κύριος Φως. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σήμερα εκπροσωπώ την ε, σκιώδη εισηγήτρια του ΕΛΚ, την κυρία Νίμπλερ, Γι' αυτό λοιπόν εξ ονόματός της θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά και εγώ τον εισηγητή για την ε, πολύ καλή δουλειά του, πολύ επικοδομητική δουλειά του σε έναν κανονισμό ο οποίος είναι αρκετά επίμαχος. Θα ήθελε όμως η κυρία Νίμπλερ να κάνει κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τα πιο ε, αμφιλεγόμενα σημεία και θα υποβάλει τις αντίστοιχες ε, τροπολογίες. Δεν θα εκπλήξει κανέναν σας ε, ότι η κυρία Νίμπλερ συνεχίζει να θεωρεί πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την παρούσα μορφή της είναι ε, χαρακτηρισμένη από υπερβολές και επαναλήψεις. Δεν Πιστεύει λοιπόν πως χρειάζονται όλες ε, αυτές και πρέπει να κρατήσουμε τα αναγκαία στοιχεία σε αυτόν τον ε, κανονισμό. Η χρήση της αρχής της χώρας προέλευσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ πρέπει να μην ξεχνάμε τον παράγοντα χρόνο Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερα στις ε, εκπομπές που αφορούν ειδήσει και τις ενομοιωτικές εκπομπές να αποφασιστεί γρήγορα το ποιος έχει τα πνευματικά δικαιώματα, να υπάρξει ρύθμιση σε αυτό. Θα ήθελε λοιπόν να ζητήσει και την στήριξή για τις σχετικές τροπολογίες, ε, οι οποίες έχουν ήδη ψηφιστεί στην Αρμόδια Επιτροπή, την Ήτρε. Επίσης, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής είναι ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την κυρία Νίμπλερ. Υπάρχουν οι αντίστοιχε τροπολογίε 191 ε, έως 200, όπου αναφέρεται, αναφέρονται τα σχετικά. επίσης, Οι 274-286 τροπολογίες αφορούν το άρθρο 3 και ε, έχουν να κάνουν με μία αλλαγή ε, στην ε, νομική βάση. Η κυρία Νίμπλερ θεωρεί πως βρίσκεται σε κίνδυνο το εφιστάμενο σύστημα, πως με την παρούσα διατύπωση κινδυνεύουν οι πιο αδύναμοι φορείς και θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει εκ των προτέρων για ε, την πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με όλους τους σκιώδες εισηγητές τι εβδομάδε που έρχονται. Και τώρα, αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ κάποια σχόλια ε, δικά μου προσωπικά, θα ήθελα να πω ότι σε γενικές γραμμές πιστεύω πως σε ένα τόσο επίμαχο θέμα όπως αυτήν την οδηγία να δούμε ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο σε ό,τι αφορά τις ε, άδειες και το θέμα της ευθύνης. Αλλά να προσέξουμε, διότι αυτά τα θέματα είναι ε, δύσκολα και είναι πολύ εύκολο να υπερβούμε τα όρια. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να παραμείνει περιορισμένο και να υπάρξει μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα στους ε, ιδιωτικούς και στους ε, δημόσιους φορείς. Μετά, να πω επίσης ότι συνεχίζω να έχω την αίσθηση πως το πεδίο εφαρμογής πρέπει να μείνει όσο το δυνατόν μικρότερο. Ιδιαίτερα, μάλιστα, δεδομένου ότι και στην Επιτροπή Πολιτισμού συμφωνήθηκε να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής. Αυτό θα ήταν καλό να το λάβετε υπόψη. Και πιστεύω πως χρειάζεται να δούμε με μεγάλη προσοχή αυτό το θέμα των δημόσιων και των ε, ιδιωτικών οργανισμών οι οποίοι ακολουθούν διαφορετικά ε, συστήματα χρηματοδότησης και χρειάζεται προσοχή λοιπόν νομικά. Μετά, ε, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε το, τη σημασία των ε, συμβάσεων για τα αποκλειστικά δικαιώματα. Η κυρία Ρέντα ήδη αναφέρθηκε ε, σε αυτά. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή και νομίζω πως ο κανονισμός κάψα πρέπει να είναι στο μυαλό μας ιδιαίτερα όταν θα επεξεργαστούμε το σημείο 5α. Ευχαριστώ κυρία Αντινόλφη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του τώρα και για την αντίδραση του που είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε τις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Είμαι πεπισμένη ότι αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά, όπω επανειλημμένω έχει δηλώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ίδιο ο πρόεδρο τη, ο κ. Γιούνκερ, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την κίνηση του να καταργήσουμε όλα τα σύνορα και όλου του γεωγραφικού αποκλεισμού, αυτέ τι πρακτικέ, οι οποίε επιτρέπουν σε ορισμένου φορεί να τεμαχίσουν με τεχνητό τρόπο την αγορά και να έχουν μεταξύ του ανταγωνισμό με αρνητικέ συνέπειε για του πολίτε. Ο κανονισμός αυτός που θέλει να διευρύνει την αρχή της προέλευσης ακόμα και στις τηλε, τηλεοπτικοακουστικές ε, μεταδόσεις online είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματική ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό θα πρέπει ταχύρυθμα να περάσουμε στην έγκριση αυτής της νομοθετικής πρότασης χωρίς να χάσουμε άλλο πολύτιμο χρόνο, ώστε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών για να περάσουμε στην ουσία της πρότασης του κανονισμού. Πιστεύω ότι η πρόταση του εισηγητή να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού ε, είναι πολύ σωστή. Τη συμμερίζουμε και πάει στη σωστή κατεύθυνση. Η προσέγγιση αυτή θα επέτρεπε όχι μόνο να εκμεταλλευτούμε τι νέε τεχνολογικέ λύσει με τα ωφέλη που προσφέρουν στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά και να διευθετήσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μια σειρά από φαινόμενα που ε, θα αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο και θα προκύψουν στην αγορά. Και να αποφύγουμε το ε, φαινόμενο της άτακτης ε, ε, διευθέτησης ε, των τεχνολογικών εξέλιξεων. Γι' αυτό έχω βάλει και εγώ κάποιες τροπολογίες για τις επιγραμμικές υπηρεσίες που αφορά, αφορά τις υπηρεσίες μόνο επιγραμμικός, δηλαδή διδακτυακός. Επίσης, η επαναμετάδοση των προγραμμάτων του ανοιχτού ίντερνετ, κάτι που θα μας επιτρέπει να ορίζουμε τον αριθμό των χρηστών χωρίς να απαιτεί είτε η χρήση τεχνολογικών λύσεων κλειστού δικτύου. Και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι θα δημιουργείται ένα control environment, όπως λέγεται, ελεγχόμενο περιβάλλον, όπου όλοι οι χρήστε θα πρέπει να έχουν κάποια είδου συμμετοχή χωρί αναγκαστικά να υπάρχει και χρηματική, χρηματικό αντίτιμο. Αυτή τη στιγμή τα προσωπικά μα δεδομένα συγκεντρώνονται αλλά με τρόπο ανώνυμο και θα πρέπει αυτό να αναγνωριστεί. Σε ό,τι αφορά την direct injection, νομίζω ότι η καλύτερη στρατηγική είναι να, ζητήσουμε, να δούμε την εφαρμογή του κανονισμού και μετά να γίνει μια ε, μελέτη αντικτύπου πιο συγκεκριμένη για να δούμε αν θα χρειαστεί σε δεύτερη φάση κι άλλη νομοθετική παρέμβαση ή όχι. Και δύο λόγια για την δυνατότητα να προβλεφθεί το α, αναντήρητο δικαίωμα στην ανταμοιβή των πνευματικών δημιουργών. Παρόλο που είμαι υπέρ τη προστασία των πνευματικών δημιουργών, νομίζω ότι η πρόβλεψη τέτοιου δικαιώματο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι ωφέλει, διότι πάνω από όλα θα προστατεύσει τους καλλιτέχνες και τους ήδη γνωστούς δημιουργούς. Θα δημιουργήσει μια σειρά από νομοθετικές επιπλοκές και δεν θα μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τις ελεύθερες πλατφόρμες όπως το Creative Commons ε, και άλλα στοιχεία που ανήκουν στο δημόσιο χώρο. αν προβλέψουμε τέτοιο δικαίωμα σε αυτόν τον κανονισμό θα είναι εσφαλμένη η κίνησή μας ε, μιας και θέλουμε να δώσουμε άλλη προστασία στο, copyright από αυτήν. Αναντήρητα είναι τα θεμελιώδη και προσωπικότατα δικαιώματα όπως το δικαίωμα του δημιουργού. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ζήτητο δικαίωμα αμοιβή ε, για την καλλιτεχνική δραστηριότητα η οποία δεν είναι πάντοτε κάτι που ξεκινάει για την ΕΣΑΗ e εκμετάλλευση και καταβολή χρηματικού αντιτίμου για το έργο που παράγει κάποιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, προσβλέπω στην αγαστή συνεργασία με τον εισηγητή και σε όλους για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Φως, θέλετε να απαντήσετε γρήγορα, ελπίζω. Θα ήθελα να επαναλάβω και να ασχοληθώ ξανά με ένα σημείο που έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση και τις σχετικές τροπολογίες για τη διαμεσολάβηση. Καταρχάς, η διαφοροποίηση στο σημείο 2, στο δεύτερο κομμάτι του κανονισμού, είναι δυνατή. Ακριβώς εάν γίνει ο διαχωρισμός ε, δημοσίου και ιδιωτικού και αν συγκρίνουμε ε, τα δύο. Το σημαντικό είναι οι παραγωγές να είναι διαθέσιμες είτε να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Πρέπει λοιπόν εδώ να είμαστε προσεκτικοί και να επεξεργαστούμε το θέμα διαφορετικά ε, από τη τη χρηματοδότηση. Εκεί τα συμφέροντα ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους νομίζω πως μπορούμε να τα συγκρίνουμε πολύ πιο εύκολα. Τώρα σε ό,τι αφορά τη διαμεσολάβηση υπάρχουν τροπολογίες με προτάσεις γι' αυτό, οι οποίες όμως για μένα βρίσκονται εκτός ε, περιεχομένου. Έχει, αναφέρονται σε νομικά ζητήματα. Η κυρία Νίμπλερ με ενημέρωσε λίγο πιο πριν για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα του χρόνου. Ε, με την υφιστάμενη πρόταση λοιπόν αυξάνεται ο, το κόστος, αυξάνεται ο χρόνος αναμονής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γεωγραφικό αποκλεισμό, επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η διαμεσολάβηση ακούγεται πάρα πολύ ωραία ιδέα, όμως είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία και μπορεί να οδηγήσει σε ε, προβλήματα παρά σε λύση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη χρήση της διαμεσολάβησης ως λύση. σας χαρακτηρίζει ούτως ή άλλως ε, η επιφυλακτικότητα κύριε Φως η κυρία Χάνιμπαλ έχει το λόγο ευχαριστώ θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά δεν είναι εύκολος ο φάκελος αυτός θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω κάποια γενικά σχόλια για τα εμπόδια και την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά Βεβαίως θέλουμε ενιαία ψηφιακή αγορά. Και δεν θέλουμε να δημιουργούμε εμπόδια όταν δεν χρειάζονται. Όμως, αυτοί που παράγουν το περιεχόμενο αυτή τη στιγμή, όποιο είναι αυτό, πρέπει να αμείβονται. Αξιοπρεπώς. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να οδηγεί σε παραγωγή ε, προϊόντων που να είναι ποιοτικά και ο καταναλωτής να μπορεί να έχει πρόσβαση σε προγράμματα και σε πληροφορίες ε, που θέλει και αξίζει. Αυτό, αυτό πρέπει να είναι το σημείο αφιτηρίας. Όσοι λοιπόν παράγουν οπτικοακουστικό υλικό ε, θα πρέπει να αμείβονται αξιοπρεπώς και θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ρύθμιση το διαδίκτυο δεν είναι απλώς κάτι το οποίο είναι ανοιχτό σε όλους και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει ή δεν θα έπρεπε να είναι εν πάση γιατί αν συμβεί αυτό τότε φτάνουμε σε παράδειγμα καταστάσεις χρειαζόμαστε ένα δίκτυο που να είναι στην υπηρεσία όλων να έχει μια συγκεκριμένη μορφή, να έχει ένα πλαίσιο και όσοι συμμετέχουν σε αυτό ε, να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες. Αυτή που να είναι η προσέγγιση μας γενικότερα για την ενιαία ψηφιακή αγορά και τη σχετική νομοθεσία. Η έκθεση το κάνει αυτό βέβαια, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω. Η γεωγραφική φραγή, το geo-blocking, είναι ένα θέμα το οποίο το βρίσκουμε συχνά μπροστά μας, είναι δύσκολο προς επίλυση. Νομίζω ότι είχαμε βρει ένα καλό σημείο ισορροπίας μετά από τις συζητήσεις που είχαμε. Εμένα με αφορά ιδιαίτερα το θέμα. Ε, το BBC, παραδείγματος χάρη, ε, εφαρμόζει το geo-blocking. Γιατί, διότι είναι δημόσια τηλεόραση, ραδιοφωνία που πληρώνεται από τους Βρετανούς. Ε, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να, να εξεταστούν. Μην το υποτιμούμε αυτό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα ζητήματα έχουν επιμέρους δυσκολίες. Δεν ξεκινάμε από το πουθενά, ξεκινάμε από ένα υπάρχον πλαίσιο. Είναι κάτι που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η αρχή της αποκλειστικότητας της εδαφικής να μπορέσει να διαφυλαχθεί σε ό,τι αφορά την πώληση προϊόντων και έργων ε, η χώρα προέλευσης. Οι εταιρείες οι οποίες παράγουν προγράμματα ντοκιμαντέρ, σειρές, ε, το κάνουν αυτό γνωρίζοντας ότι θα το πωλήσουν κατά αποκλειστικότητα σε κάποιο ε, ε, κανάλι. Ιδάλλως ε, καταραίει το πρόγραμμα και αυτό δεν θα οδηγήσει σε ένα ελεύθερο ίντερνετ το οποίο ε, θα το χαιρόμαστε όλοι. Όχι. Θα χάσουμε το περιεχόμενο αυτό, το δημιουργικό περιεχόμενο. Χρειάζεται λοιπόν εδαφική αποκλειστικότητα έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε καλά προγράμματα, προγράμματα που θέλει να δει ο κόσμος και οι καλλιτέχνες και η παραγωγή να πληρώνουν αξιοπρεπώς. Πολλά από αυτά που λέμε όταν συζητούμε για το διαδίκτυο σχετίζονται με την αμοιβή των ανθρώπων αυτών. Εάν δεν βρεθούν τρόποι για την αμοιβή των ανθρώπων αυτών που παράγουν και που δημιουργούν, ε, δεν θα υπάρχει πια το περιεχόμενο. Θέλουμε να λειτουργήσει βεβαίως ε, αυτή η αγορά με την κατάλληλη αμοιβή για τους δημιουργούς. Αυτή πρέπει να είναι βασική αρχή που θα πρέπει να διέπει τη συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω ε, αυτό που έχει κάνει ε, ο εισηγητής για το digital injection για την απευθείας διαβίβαση ε, και βεβαίως πτήθηκε το θέμα των ψευδών ειδήσεων, των fake news. Ε, fake news προκύπτουν όταν ο καθένας λέει ό,τι θέλει και λέει ότι είναι η αλήθεια. Δημοσίως. Εάν λοιπόν επιτρέψουμε υπερβολική πρόσβαση, υπερβολική χρήση χωρίς κατάλληλους διάβλους και τρόπους ε, λειτουργίας, αυτό όχι μόνο ρίνει τις ψευδείς ειδήσει, αλλά και πολλά άλλα. Και θα ήταν πραγματικά ε, τραγικό να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι άνθρωποι δεν θα εμπιστεύονται αυτό που βλέπουν στο διαδίκτυο. Είναι ένα φανταστικό εργαλείο το ίντερνετ. Έχει ε, αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Και είναι καλό αυτό, αλλά θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι αξιόπιστο και να εξακολουθεί να ε, έχει μια θετική λειτουργία. Λοιπόν, καλωσορίζω τη δουλειά που έχει γίνει. Ελπίζω να έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις έτσι ώστε να δημιουργήσουμε, να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ καταναλωτών, μεταξύ δημιουργών, παραγωγών. Ε, τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι θα αμείβονται αξιοπρεπώς στον τομέα αυτών ε, και θα μείνουν ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ την κυρία Χάνιμπολ ως μέλος της Επιτροπής μας και πριν μάθω ότι θα αναλάβω εγώ την Προεδρία είχα ζητήσει και εγώ το λόγο είχα και αυτό το πρόβλημα ε, με το μάτι μου και γι' αυτό η κυρία Μπεζερό θα διαβάσει τη δική μου παρέμβαση. Ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπεζερό. Ναι, ευχαριστώ. Χαίρομαι ε, που μπορώ να σας βοηθήσω. Κύριε Σιγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ τον συγητή για τις εξηγήσεις του. Θα είμαι σύντομος, διότι θα έχουμε τον χρόνο να να, εξετά, να παρουσιάσουμε τη θέση μα στην πρώτη συνεδρία των σχεδόν εισηγητών την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Η θέση μου, η θέση του κ. Καβαντά, έτσι, είναι η εξή. Εγώ είμαι κατά τη επέκταση του πεδίου εφαρμογή του κειμένου. Είμαι κατά τη διατήρηση του άρθρου 2 σε ό,τι αφορά την αρχή τη χώρα προέλευση, τουλάχιστον όπω προτείνεται, διότι διακυβεύει την αρχή τη εδαφικότητα των πνευματικών δικαιωμάτων. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση επί τη βάση της τροπολογίας 250 την οποία επέβαλα. Η υποχρεωτική ε, συλλογική διαχείριση πρέπει να αφορά την αναμετάδοση, την πλήρη και την ζωντανή. Ε, συμφωνώ επίσης ε, με την απευθείας σύνδεση εφόσον έχουμε ανοιχτό, ανοιχτό διαδίκτυο και κλειστό δίκτυο IP εφόσον είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των χρηστών ε, που είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι χρήστες ή που έχουν ε, κάποια συνδρομή. Ε, επίσης πρέπει να υπάρχει περαιτέρω αμοιβή για τους δημιουργούς. Είμαι κατά του forum shopping που οδηγεί σε μια εξίσωση προς τα κάτω των πνευματικών δικαιωμάτων. Ελπίζω οι συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να φανούμε σοβαροί, να μην προτρέξουμε, να ψηφίσουμε ένα κείμενο το οποίο δεν θα έχουμε εξετάσει επαρκώ τη διαπραγμάτευση. Ο κ. Καβαντά, σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και θα ήθελα και εγώ με την, για μένα πλέον να πω, προσωπική μου άποψη, ότι ε, σε τέτοιου είδου κείμενα ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η προστασία των καλλιτεχνών, των δημιουργών περνάει από την προστασία όχι μόνο των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και του ε, ε ηθικού δικαίου των ε, δημιουργών. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή Τίμο Βέλκεν για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Είναι, ήταν φανταστική η συνεργασία μας μέχρι τώρα. Και ε, θα ήθελα τώρα να πω δύο λόγια για τις κυριότερες τροπολογίες. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τη χώρα προέλευσης. Οι προτινόμενες τροπολογίες πηγαίνουν σε αντίθετη κατεύθυνση από την πρότασή μας. Κάποιες διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής ε, των υπηρεσιών σχετικά με τη χώρα προέλευσης, κάποιες άλλες προτείνουν να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής ή ακόμα και να διαγραφεί αυτό το σημείο. Να επενθυμίσω ότι η χώρα προέλευσης για μας είναι βασικό στοιχείο για τους στόχους του κανονισμού, δηλαδή να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση διασυνοριακή, πιο ανοιχτή στην ε, μεγάλη πολιτισμική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπάμε λοιπόν πάρα πολύ αυτήν την αρχή της χώρας προέλευσης. Επίσης υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που περιορίζουν την ε, ελευθερία των συμβάσεων. Θα ήθελα να πω ότι ο κανονισμός δεν αφαιρεί τη δυνατότητα χορήγησης εδαφικών αδειών. Πάντα ήταν στόχος μας να διασφαλίζεται η ε, ελευθερία των συμβαλόμενων μέρων στα πλαίσια της ε, συνθήκης τουλάχιστον. Τώρα συμφωνώ με το σημείο που είπε η κυρία Αντινόλφη η χώρα προέλευσης και αυτή η αρχή δεν θα πρέπει να αφαιρεί τη δυνατότητα ε, να έχουν ικανοποιητικέ απολαβές οι δικαιούχοι και κάτοχοι των δικαιωμάτων. Φυσικά χρειάζεται να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες, οι πληρωμές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλο το εύρος των ε, υπηρεσιών και των επιγραμμικών. Τώρα, επί, δεν είμαστε πεπισμένοι με αυτήν την δίκαιη αμοιβή, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτή εφαρμόζεται στη χώρα προέλευσης. Δεν είναι ο τρόπος δηλαδή που ο τρόπος που δίνεις μια άδεια, είναι ο τρόπος που εκμεταλλεύεσαι ε, τα δικαιώματά σου. Αυτό λοιπόν νομίζω πως... Ε, βάζει σε κίνδυνο την, τον κανονισμό και κινδεύει να περιπλέξει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Όπως γνωρίζετε αυτός ο κανονισμός είναι κομμάτι μιας, άλλη ε, πρόταση άλλης πρότασης για τα ε, πνευματικά δικαιώματα και τον εξυγχρονισμό τους. Τώρα, αναμεταδόσεις. Πρώτον, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που ε, ζητούν να καλύπτονται όλες οι OTT αναμεταδόσεις στην πρότασή μας λοιπόν έχουμε αποκλείσει τις, ε, μεταδόσεις, ε, τις ανοιχτές μεταδόσεις στο διαδίκτυο. Καταρχάς γιατί αυτές οι υπηρεσίες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, οικονομικά ε, και μη. Μετά δεν συνδέονται με κάποια συγκεκριμένη υποδομή. Και τρίτον, για να υπάρχει έλεγχος πρέπει να είναι ελεγχόμενο και το, ελεγχόμενο και το περιβάλλον. Σε ένα ανοιχτό ε, διαδίκτυο δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν οι σχετικοί κίνδυνοι. Απ' την άλλη, υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που ζητούν να διαγραφεί από το άρθρο 3, από το πεδίο εφαρμογή, ε, το σημείο για τις υπηρεσίες μετάδοσης από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί, διότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι κλειστά δίκτυα. Γι' αυτό θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα τους λόγους πίσω από αυτήν την διαφοροποίηση και, τον, ε, και την εξαίρεση αυτών των ε, υπηρεσιών. Μετά, για τις απευθείας διαβιβάσεις, υπάρχουν όντως αυτές οι τροπολογίες που ζητούν ε, επανεξέταση των διατάξεων. Αυτό δεν ε, καλύπτεται προς το παρόν από την πρόταση της Επιτροπής. Οι απευθείας διαβιβάσεις είναι κάτι πολύ περίπλοκο, όχι μόνο νομικά, αλλά λόγω των συμβατικών υποχρεώσεων που μπορούν να είναι πολλές και διάφορες, είναι και πρακτικά δύσκολη. Το δικαστήριο στην ε, περίφημη απόφαση SPS Σάμπαμ απεφάνθη όπως ε, αναγνωρίζεται η ανάγκη ανάλυσης ε, κατά περίπτωση. Οι απευθείας διαβιβάσεις όσο γνωρίζουμε χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή μόνο σε εθνικά ε, πλαίσια και οι τέτοιες ε, μεταδόσεις ε, είναι ελάχιστες. Δύο μόνο τέτοιες χώρες αντιμετωπίζουν θέμα, το Βέλγιο και οι κάτω χώρες με τις απευθείας διαβιβάσεις. Το Βέλγιο πρόσφατα βρήκε μια λύση στο πρόβλημα μετά από μακρόχρονες και δύσκολες διαβουλεύσεις. Νομίζω πως λοιπόν θα είναι πολύ διστακτικοί και δεν θα αλλάξουν θέση τόσο εύκολα θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό πρώτον να γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης, να ζυγίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα υπέρ και τα κατά. Δεν είμαι πεπισμένο ότι υπάρχουν πιο πολλά υπέρ από ό,τι κατά με την εισαγωγή αυτού του μέτρου. Νομίζω μάλιστα πως θα προσθέσει ακόμα περισσότερες ε, δυσκολίες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα χαρώ πολύ να συνεισφέρω στην ε, συζήτηση με τη δική μου εμπειρία. Ευχαριστούμε. Κλείνει λοιπόν το, η συζήτηση για το σημείο αυτό. Περνάμε στο σημείο 18 τώρα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φως. 468, 468 είναι ε, Αγαπητέ Άξελ, παρακαλώ να είσαι όσο γίνεται πιο σύντομος, διότι όπως ξέρετε δεν έχουμε συνεδρία στο απόγευμα. Ε, κανένα από τα σημεία του πρωινού δεν μπορεί να εξεταστεί στο απόγευμα. Οπότε στα 58 λεπτά που μας μένουν καλό θα είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε το, θέ, το σύνολο της μέρες διάταξης. Θα να ολοκληρώσουμε. Κύριος Φως. Σας ευχαριστώ πολύ. 470 τροπολογίες υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Γιούρι. Η θέση μου είναι λίγο πολύ γνωστή. Αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καταστροφική και θα είναι καταστροφική μάλλον μέσω πρόθεσμα ε, σε ό,τι αφορά τη σχέση της με τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων. Λίγο πολύ νομίζω πως αγνοήσαμε ότι υπάρχει και ένας άλλος κανονισμός. Οι χρήστες Νομίζω πως ε, με την παρούσα πρόταση δεν, δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα πια. Γιατί πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί κανονισμοί, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να διέπονται από δύο διαφορετικά ε, συστήματα. Δεν, ξέρουν, δεν θα ξέρουν τι συμβαίνει. Τώρα υπάρχει υπερβολική ρύθμιση, υπάρχει προσκόλληση σε παλιές δομές τις οποίες διατηρούμε. Να σας υπενθυμίσω πως υπάρχει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ε, με τον οποίο υπάρχουν έντονες αντιθέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, με τα cookies για παράδειγμα. Ε, και εάν θέλουμε να ενισχύσουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία των δεδομένων με αυτήν την πρόταση θα κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Θεωρώ πως ε, πρέπει να υπάρχει συμφωνία αυτή τη πρόταση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, ιδιαίτερα των ε, προσωπικών δεδομένων. Δεν υπάρχει τώρα μεγάλη ασάφεια σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Δεν ξέρει κανείς σε ποιο καθεστώς ε, υφίσταται. Μετά υπάρχουν και τα μεταδεδομένα και το ζήτημα της ε, σύμφωνης γνώμης. Νομίζω πως ε, αυτή τη στιγμή έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από το αρχικό σκεπτικό ώστε υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Πολλές φορές δεν ζητείται η συγκατάθεση ή μάλλον ε, πολλές φορές ε, όταν ζητείται συγκατάθεση και το κείμενο πρέπει να διαβάσει κανείς είναι πάρα πολλών σελίδων, δεν το διαβάζει καν και απλά δίνει τη συγκατάθεσή του χωρίς ε, δεύτερη σκέψη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα μετά ε, με, το, με τη διαχείριση αυτών των δεδομένων. Εδώ πέρα πέφτουν, ε, εδώ πέρα υπάρχουν και θέματα marketing. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που αφορούν από τα cookies μέχρι και κατάργηση ολόκληρων κεφαλαίων. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως έχουμε πολλή δουλειά ακόμα για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για την διεξοδική σας ε, και σύντομη παρουσίαση. Η κυρία Κότμαν. Ο... Η κυρία Κότμαν έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Ντεβό, ζητά συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, οπότε μου ζήτησε να διαβάσω. Τις απόψεις της Ευχαριστεί τον εισηγητή και τους κοιόδες για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την ενέργεια που έχουν καταβάλει για να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα. 468-470 τροπολογίες για μια γνωμοδότηση δεν είναι και λίγο. Οι συνάδελφοι της ΛΥΜΠΕ ήδη διαπραγματεύονται τις συμβαστικέ λύσεις και σκοπεύουν να ψηφίσουν στις 11 Οκτωβρίου. Φαίνεται να μην έχουμε πολύ χρόνο για περαιτέρω συζητήσεις. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι όπως ξέρετε εμείς ως ομάδα δεν ε, συμφωνούμε με τη γραμμή του κυρίου Φως. Θεωρούμε ότι ο κανονισμός αυτός είναι αναγκαίος, θα συμπληρώσει τους ειδικού νόμους για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το GDPR. Τον κανονισμό δηλαδή για την γενική προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Θα ε, προστατεύσει τους πολίτες παρέχοντας περισσότερες υπηρεσίες Όπω λέει η κυρία Ντεβό, όπω διαβάζω και από τι τροπολογίε τη, οι συνάδελφοι από άλλε ομάδε, άλλοι Πράσινου και Γκουέ, συμμερίζονται και εκείνη τη δική μα άποψη. Ελπίζω λοιπόν ότι ο κύριο Φω θα το λάβει υπόψη. Πρέπει να βρούμε κάποιε συμβαστικέ λύσει σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Άντερσον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θα είμαι σύντομος. Η πράσινη είναι κατά κύριο λόγο υπέρ της πρότασης της Επιτροπής και, κατά αυτήν, και σε αυτή την κατεύθυνση θα ψηφίσουν και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ως εκπρόσωπος της ομάδας μου ανυπομονώ για τις τροπολογίες τις οποίες ελπίζω να δω αλλά ανησυχώ λίγο για το χρονοδιάγραμμα. Εάν θα έχουμε χρόνο να τις μελετήσουμε τις 468 τροπολογίες πριν την ψηφοφορία μας, αλλά ανυπομονώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ντινόλφη. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπημένοι μου συνάδελφοι και εγώ θέλω να εκφράσω κάποιες απόψεις ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άποψη της privacy του ιδιωτικού βίου σε ηλεκτρονικό, στο ηλεκτρονικό επίπεδο έχει πολύ γενική και προηγμένη νομοθεσία σε σχέση με άλλες ε, χώρες του δυτικού κόσμου. Όμως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ήθελα λοιπόν να πω τα εξή. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του εισηγητή για το γεγονός ότι η έκθεση αυτή αναφέρεται στο νέο τηλε, κώδικα για τι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε που ακόμη δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Υπάρχει λοιπόν αβεβαιότητα για ορισμένα σημεία. Κατανοούμε, αλλά δεν συμμεριζόμαστε τι ε, παρατηρήσεις ότι είναι λέξ σπετσιάλη, ειδικό νομοθέτημα ε, η πρόταση αυτή για την προστασία των ηλεκτρονικών ε, δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων. Και αυτό γιατί οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες έχουν τέτοιε ιδιαιτερότητες, τόσο περιπλοκές, που θα πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε με πολύ ειδικότερε διατάξεις που να υπερισχύουν των γενικών. Υπό αυτήν την έννοια θα προτείνουμε τροπολογίες γιατί θεωρούμε ότι μπορεί το πεδίο της οδηγίας να καλύπτει όχι μόνο τη ροή των ε, δεδομένων από τις ε, ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή των τηλεφωνημάτων, των μηνυμάτων WhatsApp και άλλων μορφών ψηφιακής επικοινωνίας αλλά και τα μεταδεδομένα. Αυτά τα οποία πολλές φορές ε, τηρούν οι πάροχοι των υπηρεσιών. Ε, δεδομένα που βρίσκονται στο διαδίκτυο και στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Ε, θα πρέπει λοιπόν να στρέψουμε την προσοχή μας και στις διεθνείς μας συμφωνίες και την προστασία των δεδομένων που ε, αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργώντας μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των θεωριών για την προστασία των δεδομένων και το τι κυκλοφορεί για τους πολίτες μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι μεγαλύτεροι εμπειρογνώμονες της ηλεκτρονικής ασφάλειας πρόσφατα ε, σε μια συνέντευξη ε, λέγαν ότι στην αρχή θεωρούσαν ότι το Google λόγω των δεδομένων που συγκεντρώνει από τις αναζητήσεις μου με γνωρίζει καλύτερα και από τη γυναίκα μου. Η αλήθεια είναι ότι το Google έχει καταφέρει να με γνωρίζει καλύτερα από μένα τον ίδιο, διότι ξέρει για μένα πράγματα που δεν τα ξέρει τη γυναίκα μου. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που μας περιμένει λοιπόν. Αυτό ήθελα να πω με, αυτήν την, ε, ε, με αυτό το παράθεμα και ελπίζω να έχουμε μια πρόσφορη και αποτελεσματική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Αλλά από μένα θα την παρουσιάσει η κυρία Μπερζερό. Κύριε ε, εισηγητά, αγαπητέ Άξελ, κύριοι συνάδελφοι, είναι θεμητό να θέλει κανεί να εφαρμόσει του κανόνε αυτού του κανονισμού βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων. Βρίσκω ότι το κείμενο τη Επιτροπή πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση και είναι ε, δουλειά του Κοινοβουλίου να το συμπληρώσει. Είναι σημαντικό το κείμενο αυτό να μην αντιφάσκει με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 11, είναι σημαντικό το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερισχύσει του εθνικού εκτός από τις περιπτώσεις με συγχωρείτε εκτός από τις περιπτώσεις διαφύλαξης της ε, ασφάλειας ή της άμυνας των κρατών. Θεωρώ ότι ε, όλες οι περιπτώσεις χρήσης cookies δεν πρέπει να ε, απορριφθούν, αλλά θα πρέπει να επαναπλησιώσουμε τη χρήση του χρήση τους. Επίσης οι παράμετροι απορρίτου και προστασίας του ιδιωτικού βίου πρέπει να πλαισιωθούν σωστά ώστε οι τελικοί χρήστες να μπορούν να αντιταχθούν στην λήψη ε, επικοινωνιών και την τήρηση των δεδομένων χωρίς να υπάρχει συγκατάθεση θα συμμετάσχω στην ε, εκπόνηση τη έκθεση με την υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ε, η Επιτροπή δεν έχει ζητήσει το λόγο. Όντω, ωραία. Ε, προχωρούμε στο επόμενο σημείο. Με βολεύει αυτό γιατί έχουμε καθυστέρηση. Επόμενο σημείο στην εμμύρια διάταξη. Σα ευχαριστώ. Επόμενο λοιπόν σημείο στην εμμύρια διάταξη. Σημείο 8. Εκ, ε, παρουσίαση. Ο κύριος Φως. Μια και ανέλαβε. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ και τον Πάβελ Σβόμποντα σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να διαβάσω κάποιες από τις προτάσεις του. Αγαπητοί συνάδελφοι, μου ζητήθηκε από τον πρόεδρο να παρουσιάσω λοιπόν εκ μέρους του ε, κ. Τσαμπάσκη κάποιες σκέψεις για την πρόταση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση της δέσμευσης και δίμευσης και θα διαβάσω λοιπόν το σύντομο σημείωμα που μου έδωσε. Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας στη σημερινή εποχή, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να εντοπίσουμε ε, περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε επικράτη άλλου κράτους μέλους μέσω μιας αποτελεσματικής διαδικασίας κατάσχεσης. Αυτό το, αυτός ο χώρος του ποινικού δικαίου είναι ιδιαίτερα κατακαιρματισμένος λόγω των διαφορών ε, στις, ε, στα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Υπάρχει λοιπόν μια πληθώρα προσεγγίσεων νομικών στα θέματα αυτά. Στο, στην 3, στο κανονισμό 3 Απριλίου για τη δέσμευση και βήμευση περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια ποινικών ερευνών προσπαθούμε να ε, θεσπίσουμε ελάχιστους κοινού κανόνες σχετικά με τα μέτρα κατάσχεσης. Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας ήταν Οκτώβριο του 2016. Ωστόσο, προτού διαβάσουμε την ε, αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα δημοσιευτεί το τέλος του 2018, έγινε προφανές ότι ακόμα και στην καλύτερη των περιπτώσεων η νέα οδηγία είναι μόνο ένα μικρό βήμα προς την περαιτέρω ευθυγράμμιση των κανόνων σχετικά με την ε, κατάσχεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο μετά, ε, ακριβώς μετά την... Ε, εξέταση της οδηγίας ε, προσπάθησε να κάνει μία ε, ενδελεχή έρευνα για τους κανόνες ε, περιθέσμευσης και δίμευσης. Στα πλαίσια λοιπόν της πρότασης αυτής θα ήθελα να την καλωσορίσω και να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυξημένη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του εντοπισμού, της ε, δέσμευσης ε, και της ε, διήμευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Η αμοιβαία αναγνώριση είναι πάρα πολύ σημαντική στα πλαίσια της δικαστικής συνεργασίας και πρέπει να παραδεχτώ ότι η επιλογή κανονισμού αντί για μια απόφαση πλαίσιο ή αντί για μια οδηγία είναι μια πολύ καλή είδηση που θα δημιουργήσει περισσότερη ομοιογένεια στην λειτουργία στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και θα αποφύγει κερματισμούς που θα δυσχεράνουν την ε, προσπάθειά μας για τη μετώπιση αυτού του ε, φαινομένου. Η πρόταση λοιπόν εισαγεί διάφορους ε, λόγους άρνησης της εντολής δέσμευσης και διήμευσης σε περίπτωση που τα νομικά συστήματα δεν επαρκού, των κρατών μελών δεν επαρκούν. Χωρίς φυσικά να ε, θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα έτσι όπως αυτά αναγράφονται στην ε, Χάρτα των Θεμελιώδων Δικαιωμάτων και στην Θήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν να βελτιώσουμε περαιτέρω την... Ε, ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, να γίνει πιο γρήγορη συνεργασία αυτή, να υπάρχει διαθεσιμότητα πληροφοριών, να υπάρχει γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών και αυτό θα διασφαλιστεί μέρη και από τα σύγχρονα συστήματα, υπολογιστικά συστήματα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει σαφήνεια ε, σε ό,τι αφορά την ε, συμμόρφωση του, ε, της πρότασης αυτής με τους ε, υπάρχοντες κανονισμούς, αλλά και είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η υποχρέωση ενημέρωσης και κοινοποίηση σε περίπτωση ε, δέσμευσης ε, περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να, έχετε να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίηση όλων των ε, καταλήλων ένδικων μέσων. Είναι πολύ σημαντικό να πληροφορείτε και ο κάτοχος λοιπόν των περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεσμεύονται. Να σας υπενθυμίσω πως στις 12 Σεπτεμβρίου έχουμε την προθεσμία υποβολής τροπολογιών και η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 10 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φως. Κυρία Κάφμαν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ας αναλογιστούμε τα ποσά και τα περιουσιακά στοιχεία, την κινητή και ακίνητη περιουσία που διακινείται και προέρχεται από εγκληματικέ δραστηριότητες. Σκεφτείτε πώς θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε τους εγκληματίες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να συνεχίσουν την εγκληματική τους δραστηριότητα. 98,9% των εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες ε, δεν μπορούν να κατασχεθούν. Αυτά συνδέονται μετά και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες και φαίνεται πως υπάρχει μια προφανής ανάγκη βελτίωσης της νομοθεσίας εδώ. Όπως και ο εισηγητής, έτσι και εγώ στηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πρόταση κανονισμού, έτσι ώστε να απλουστευθεί σημαντικά το νομικό πλαίσιο η πρόταση που έχουμε αυτή τη στιγμή δίνει κάποιες ε, περαιτέρω διευκρινήσεις σε ορισμένα σε και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Θέλω να σταθώ κι εγώ σε ένα-δυο σημεία τα οποία απασχόλησαν και τον κύριο Σφόμποντα από όσο γνωρίζω. Όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν έτοιμα ε, δέσμευσης ή δίμευσης περιουσιακών στοιχείων τότε πρέπει να λαμβάνεται ε, και μία ξεκάθαρη αιτιολόγηση γι' αυτό. Οι αρμόδιες αρχές λοιπόν των κρατών μελών φυσικά επίσης χρειάζονται σύγχρονα συστήματα ε, ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών έτσι ώστε αυτή η ανταλλαγή να γίνει ε, γρήγορα και με ασφάλεια. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για παρανόμως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία. Τώρα, μαζί με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές, ε, θα είμαι, είμαι σίγουρη πως θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ ξανά. Ευχαριστώ. Δεν φαίνεται να θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζήτησε το λόγο. Δεν αλλάζει κάτι. Κερδίζουμε και χρόνο έτσι. 12 Σεπτεμβρίου προθεσμία για την υποβολή τροπολογίων. για το θέμα αυτό ήθελα να σας πω ότι θα περάσουμε στο επόμενο. Βυρσνή Ροζιέρ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξετάζουμε αυτή τη στιγμή τις τροπολογίες 200 221 ε, τροπολογίες του σχέδιο έκθεσης από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, σχεδόν Χαιρόμαστε βέβαια που στην ευρύτερη φιλοσοφία ε, των τους ε, οι τροπολογίες υποστηρίζουν ε, σχεδόν όλες οι ομάδες την ιδέα μιας οριζόντιας νομοθεσίας που είναι και ο πρώτος στόχος αυτής της έκθεσης. Οπότε είναι πραγματικά εξαιρετικά ικανοποιητικό το γεγονός ότι όλοι ακολουθούμε λίγο πολύ την ίδια οδό, στο ίδιο πνεύμα με το σκηνούμαστε. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν και αποκλήσεις. Εξού και οι συμβαστικές προτάσεις σε μια σειρά αποζητήματα. Το πρώτο είναι ο ορισμός του whistleblower. Πολλοί, πολλές ομάδες έχουν υποβάλει τροπολογίες για να μπει η έννοια της καλής πίστης ε, στον ορισμό. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια ανησυχία την οποία όλοι συμμεριζόμαστε. Νομίζω πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει ένα διαχωρισμό μεταξύ ε, της, του συναγερμού όντω και, και τη ε, δυσφήμιση. Έτσι της λάσπης. Τώρα, η έννοια της καλής πίστης ε, ανοίγει βέβαια το δρόμο ε, στο να αρχίσουμε να αμφισβητούμε τις προθέσεις του whistleblower που ε, όταν έχουμε μέσα σε μια διαδικασία όπου υπάρχουν πολύ έντονες πιέσεις δικαστικές αυτό θα μπορούσε τελικά να αποδυναμώσει την προστασία από το whistleblower. δηλαδή να αρχίσουμε να τον κρίνουμε και ηθικά ή να ε, αναλύσουμε μέχρι εσχάτων τις προθέσεις του, ε, ούτως ή άλλως είναι σε έθραυστη θέση, διότι διώκονται οι άνθρωποι αυτοί. Οπότε εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι να βρούμε μια διατύπωση που να δείχνει ότι βεβαίως ε, ο whistleblower όταν ε, κρούει το κούρνο του κίνδυνου πρέπει να είναι βέβαιος ε, για, την, για τα στοιχεία τα οποία φέρνει, τα οποία μοιράζεται μαζί μας. Οπότε θα πρέπει να αποφύγουμε ε, βεβαίως τις διφημίσεις και τη λάσπη, αλλά ε, να βρούμε μια εναλλακτική λύση και να μιλάμε για καλή πίστη. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ε, ορισμό ε, ότι το, πεδίο μάλλον η προστασία αναφορά μόνο τις σχέσεις τις συμβατισιακές Κάποιες άλλες ομάδες όμως ε, είπαν ότι πρέπει να το διευρύνουμε αυτό και να αφορά ε, όποια και όλες τις σχέσεις, ε, οποιαδήποτε σχέση μπορεί να έχει whistleblower με, τις, ε, με τους οργανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται. Υπάρχει ένα επίκαιρο παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε το φαρμακευτικό εργαστήριο και της υπηρεσίας φαρμάκων Εκεί ο whistleblower, η κυρία Φρα, Φρασόν, δεν είχε καμία απολύτω ε, εργασιακή σχέση ούτε με την εργαστήριο Σερβιέ, ούτε με την ε, υπηρεσία φαρμάκου, αλλά αυτή είναι η οποία έξω από τον κρόνο του κινδύνου. Ε, δεν έχουμε βεβαίως πολλά τέτοια παράδειγματα, αλλά θα είναι προβληματικό μια, σε μια τέτοια περίπτωση το άτομο αυτό να μην χαίρει προστασία. Οπότε μάλλον θα ήθελα ο ορισμό να είναι και εδώ όσο γίνεται πιο ευρύ. Το άλλο ζήτημα ε, όπου υπάρχουν διαφωνίες είναι ο ορισμός του δημοσίου συμφέροντος. Η εμπασχεπτώση της ε, πώς ορίζουμε ότι πλήττεται το γενικό συμφέρον, το κοινό συμφέρον. Υπάρχει η πρόταση της έκθεσης που ε, αναφέρεται σε μια γενική αρχή και μετά έχουμε και ένα κατάλογο παραδειγμάτων που έρχονται κάπως να διανθίσουν ε, το τι εννοούμε. Ε, κάποιοι θέλουν να περιορίσουν τον κατάλογο αυτό των παραδειγμάτων. Εγώ νομίζω ότι έτσι όμως απομακρυνόμαστε από την πραγματικότητα διότι όντως ε, καταγγέλλονται κάποια πράγματα αφορούν, που αφορούν τους πολίτες ε, δύσκολο δηλαδή ε, παραδείγματος χάρη να βγάλουμε από τον κατάλογο την σύγκρουση συμφερόντων, τα θέμητα συμφέροντα. Αυτό αφορά προφανώς το γενικό συμφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα πολλοί ε, ζητούν ειδικού κανόνες για ευαίσθητου τομεί, για ευαίσθητου κλάδου ή να προστατεύσουν ρητά ε, κάποιο απόρριτο ε, που δεν αφορά οικονομικά συμφέροντα αλλά δελολογικά ή εμπιστευτικότητας. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να το σκεφτούμε, να δούμε δηλαδή, να προλέψουμε κάποιες εξαιρέσει. Ε, θα υποβάλω μια σχετική πρόταση στα πλαίσια των συμβιβασμών. Υπάρχει ένα σημαντικό σημείο ε, διαφωνίας για τον ανώνυμο χαρακτήρα. Πέρα από το σεβασμό της εμπιστευτικότητας του whistleblower, είναι πολύ σημαντικό αυτή την προστασία, ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, ανώνυμος, να, να, να, να την ανωνυμία του. ξέρουμε ότι οι πιο ευάλωτοι ε, θα αποτραπούν από το να ενημερώσουν διότι φοβούνται την έκθεση. Το να μπορέσουμε λοιπόν να πλαισιώσουμε, ε, με, πλαισιωμένο τρόπο μάλλον, να προλέψουμε ανωνυμία ε, είναι σημαντικό. Είναι σημαντική αυτή η δυνατότητα. Ένα άλλο στοιχείο στην έκθεση έχει να κάνει με τα μέσα της ε, ειδοποίησης. Είναι ένα βασικό, ένα κεντρικό σημείο της συζήτησης που θα μας απασχολήσει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ενημέρωση εντός της οργάνωσης, στις αρμόδιες αρχές ε, για να παρέμβουν και να ρυθμίσουν μια κατάσταση και στο ευρύ κοινό. Ε, βεβαίως υπάρχει μια κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις. Κάποιες ομάδες ε, θέλουν να είναι ανοιχτή η δυνατότητα να μπορεί κάποιος να δημοσιοποιήσει όπως θέλει. Κάποιοι άλλοι θέλουν εφόσον να υπάρξει ε, άμεση δημοσιοποίηση να μην υπάρχει προστασία. Ε, είμαστε στο άλλο δηλαδή άκρο. Πρέπει βεβαίως πιστεύω να υπάρχει προστασία ακόμα και όταν ο whistleblower το διαδίδει στο ευρύ κοινό. Το γεγονός το μάθαμε αυτό και με την φοροαποφυγή. Ο Αντουάν είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ε, όταν έχουμε την καταγγελία συμφωνιών ε, μεταξύ του εργοδότη, δηλαδή της οργάνωσης του θεσμού και των διοικητικών αρμόδιων αρχών, ε, τότε πού να απευθυνθεί κανείς στο εσωτερικό επίπεδο, ούτε στην κυβέρνηση του μπορεί να πάει, στις δημόσιες αρχές, ούτε στην εταιρεία του. Η μόνη λύση στην περίπτωση αυτή είναι ε, να το ε, δημοσιοποιήσει το ευρύ κοινό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, και είναι κάτι που πρέπει να προστατεύεται. Οι συζητήσεις αυτές θα συζητηθούν βέβαια, θα συνεχιστούν βέβαια. Τώρα υπάρχει το θέμα του βάρους της απόδειξης, που το οποίο με την καλή πίστη. Η προστασία στην περίπτωση κυρώσεων και αντίμετρων είναι κάτι το οποίο, στο οποίο υπάρχει μια κάποια ομοφωνία. Κάποιοι λένε ότι όχι μόνο ε, πρέπει να αποζημιωθεί ο whistleblower, αλλά θα πρέπει ε, και να επιβραβευτεί στη συνέχεια οικονομικά από το κοινωνικό σύνολο. Βέβαια αυτό μας πάει σε ένα κάπως σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι ε, δεν είναι και στην κουλτούρα μας την ευρωπαϊκή και δημιουργείται, δημιουργείται από εκεί πέρα και μία ε, καχυποψία γύρω από τα κίνητρα του whistleblower. Θα το συζητήσουμε μεταξύ χειρών εισηγητών, αλλά νομίζω ότι αυτό μας απομακρύνει ε, από, ε, το τι, από την έννοια, την ίδια την έννοια του whistleblower. Τώρα έχουμε, ε, υπάρχει το θέμα των μέσων που διαθέσουμε και υπάρχει το θέμα της νομικής βάσης. Ε, θα ανοίξουμε εδώ κάποιες Κάποιου δρόμου από εκεί πέρα η Κομισιόν ε, θα προχωρήσει με πιο συγκεκριμένο τρόπο προ την κατεύθυνση αυτή. Η πρώτη συνάντηση των σκιών εισηγητών έλαβε χώρα χθε. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του σκιών εισηγητέ από όλε τι ομάδε για τη συμμετοχή του, την ενεργή και εξαιρετικά επικοδομητική συμμετοχή του, που σίγουρα θα συνεχιστεί μια και υπάρχει άλλη μια συνάντηση λίγο πριν ψηφοφορία που προβλέπεται στι 28 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ. Μιλάτε πολύ γρήγορα, ε, για να είστε και σύντομοι βέβαια παρακαλώ και οι υπόλοιποι να κάνουν το ίδιο όσο γίνεται πιο σύντομα ε, διότι έχουμε μόλις μισή ώρα στη διάθεσή μας ε, και πρέπει να κλείσουμε όλα τα θέματα. Ο κ. Χρυσογόνος έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά της σε αυτό το θέμα. Η προστασία όσων καταγγέλουν παρατυπίες είναι, είναι προς το κοινό συμφέρον. Η αποτελεσματική προστασία τους θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα για να αποτρέψουν και να αντιμετωπίσουν ε, παραβιάσεις της ε, αρχής της ε, ακαιρεότητας που απειλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυξάνουν την ενεργία, περιορίζουν ή διαστευλώνουν τον ε, δίκαιο και ε, θέτουν σε κίνδυνο τα δημοκρατικά, ε, τους δημοκρατικούς θεσμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προστασία λοιπόν των καταγγελόντων είναι πάρα πολύ σημαντική διότι αποκαλύπτουν πληροφορίες, προωθούν την δημόσια λογοδοσία των κρατικών θεσμών και μη αποτρέπουν την ε, απάτη και τη διαφθορά, ενισχύεται η δυνατότητα ανταπόκρισης ε, και αντιμετώπισης απειλών, ωστόσο πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα έτσι ώστε να αναπτύξουμε ένα σταθερό έδαφος με ανοιχτό χαρακτήρα και ακαιρεότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να βοηθά την προστασία των ε, καταγγελόντων. Είναι κάτι που πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη και να υπάρχει εναρμόνιση. Ωστόσο δεν συμβαίνει αυτό. Μόνο ελάχιστα κράτη-μέλη έχουν ε, δημιουργήσει και έχουν θέσει σε λειτουργία αποτελεσματικά συστήματα προστασίας αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να ε, είναι προστατευμένοι έτσι ώστε να μπορούν να, να ε, κάνουν τις καταγγελίες τους. Ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας για την αποκάλυψη πληροφοριών με τη συνέπεια ενδεχομένως όσοι καταγγέλουν ε, παρατυπίες να αντιμετωπίσουν πειθαρχικά μέτρα τα οποία ξεπερνούν τις εργασιακές τους σχέσεις. Σύμφωνα με μία έρευνα του οσα πάνω από το 1 τρίτο των οργανισμών με μηχανισμούς ε, ε, καταγγελίας, δεν έχουμε, μηχανισμούς αναφοράς δεν έχουν κάποια μέτρα προστασίας των ε, όσων καταγγέλουν παρατυπίες ως αποτέλεσμα για να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εγγυάται υψηλή προστασία ε, των καταγγελόντων και στον ε, δημοτικό και στον, και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε όλα τα θεσμικά όργανα χρειάζεται μια σαφή διαδικασία για την προστασία τους αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένους ορισμούς, αποτελεσματικά ε, μέτρα προστασίας από αντίπεινα και εξαιρέσεις από ποινικές ε, και ε, μη διώξεις. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι επιχειρήσεις να έχουν ένα αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα προστασίας γιατί θεωρώ πως η, έννοια του whistleblower είναι μια έννοια που ερμηνεύεται ευρύτατα ε, ερμηνεύεται η καταγγελία ως μια πράξη που ε, υπονομεύει το κοινό συμφέρον χωρίς να υπάρχουν μαρτύρες από πρώτο χέρι. Ιδιαίτερα όσοι καταγγέλουν παρατυπίες οι οποίες αφορούν το, κοινό, το δημόσιο συμφέρον πρέπει να προστατεύονται παρκώς. Τα μέτρα που λαμβάνονται λοιπόν ε, εναντίον τους πρέπει να ε, σταματήσουν και πρέπει όσοι κάνουν τις καταγγελίες αυτές να λαμβάνουν επαρκή αποζημίωση για την ε, ζημία στην οποία μπαίνουν και για υλικές και για ηθικές ε, λοιπόν, ε, ζημιές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένας επαρκής μηχανισμός προστασίας τους και επαλήθευσης της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δίνουν. Χρειάζεται λοιπόν συγκεκριμένα δεδομένα, δείκτες, συγκριτική αξιολόγηση. Χρειάζονται ιστότοποι με εύκολη πρόσβαση σε όλη την επικράτεια της Ένωσης που θα παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την προστασία των καταγγελόντων και πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να γίνονται εκεί ε, καταγγελίες με ε, μεγάλη εμπιστευτικότητα. Μετά πρέπει να υπάρχουν διάφορα σημεία επαφής, ε, ιστοσελίδες, ιστότοποι, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Κοινοβούλια των κρατών μελών έτσι ώστε να δέχονται τις καταγγελίες από τους πολίτες και οι καταγγέλλοντες πρέπει να λαμβάνουν στήριξη και επαρκή βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τα ενδεχόμενα αντίπεινα και σε περίπτωση παράνομης συμπεριφορά. πρέπει να υπάρχει επαρκής προστασία με, όποιο, ε, με όλους τους δυνατούς τρόπους σεβόμενοι πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα υποβάλω τις σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ. Εκπρόσωπο την Ρόζα Αστερά, τη και Δησηγήτρια κυρία Εστράς θέλει να ευχαριστήσει τον ε, εισηγητή για την ε, σύνταξη του σχεδίου έκθεσης, για την προστασία των ε, πληροφοριοδοτών, των whistleblowers, ως προς την ίδια την έκθεση να θυμίσει ότι περισσότερο οι αριστερές ομάδες έχουν προωθήσει το θέμα αυτό. Παραδοσιακά το ΕΛΚ ήταν της άποψης ότι το θέμα αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και θεωρείται αρκετά επίμαχο ζήτημα. Μετά τα τελευταία σκάνδαλα, το ΕΛΚ έχει ταχθεί υπέρ της λήψη μέτρων για την προστασία των λογοδοτών, λεωφοριοδοτών, αλλά πάντοτε ως αντίβαρο των ακραίων θέσεων της αριστεράς. Τις βρίσκουμε προβολικές το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα του Συμβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να παρατηρηθεί ότι αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το εξετάσει κάποια στιγμή, παρόλο που θεωρεί ότι είναι δύσκολο να ε, γίνει έναρξη νομοθετικής διαδικασίας για την οριζόντια προστασία των πληροφοριοδοτών. μιας και δεν υπάρχει γι' αυτό νομική βάση. Ως προς το σχέδιο έκθεσης, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ε, οριζόντια νομοθετική πρόταση επί του θέματος πριν το τέλος της χρονιάς. Για το ΕΛΚ αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Δεν μοιάζει να υπάρχει σχετικά νομική βάση για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία και η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να πρετανεύσει και να γίνει σεβαστή. Θα πρέπει ο ορισμός για τους whistleblowers να ε, γίνει αποδεκτός και από την ομάδα μας, διότι αναφέρονται παράπονα στο δημόσιο και ιδιωτικό ε, τομέα. Κάποια, όπως η ανάγκη προσφυγές να βασίζονται ε, σε κίνητρα μεταξύ των οποίων και καλή πίστη, αυτά θα πρέπει να ε, εξαλειφθούν. Δεν υπάρχει τρόπος να υποβληθούν τέτοιες προσφυγές θα πρέπει η Επιτροπή να προβλέψει ένα σύστημα για την υποβολή προσφυγών και η προσφυγή πρώτα να υποβάλλεται εσωτερικώ και μετά στην αρμόδια αρχή. Αυτή η πρόταση μα βρίσκει συμφωνούσα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και οι άνθρωποι που ε, δεν ε, περνάνε από αυτέ τι διαδικασίε και πάνε απευθεία στον τύπο, θα πρέπει και αυτοί να προστατεύονται. Ένα από τα πλέον αφιλεγόμενα είναι ότι για να προστατευτούν οι πληροφοριοδότε και να ε, αναχαιτιστούν τα αντίπεινα, η δυνατότητα αντιστροφή του βάρου απόδειξη, τη υποχρέωση του βάρου απόδειξη, θα πρέπει να διατίθεται εφόσον χρειάζεται. Από νομική πλευρά για μα αυτό είναι ε, παράλογο. Ε, Επίση η ανώνυμη υποβολή στοιχείων, αυτό δεν μα αρέσει. Ευνοεί την ε, καταχρηστική χρήση των μηχανισμών και θα πρέπει να έχει κανεί υπόψη ότι ο κανονισμό φω μπορεί να βλάψει πολλού αθώου θα πρέπετε ότι μια ψευδής έκθεση μπορεί να βλάψει πολλούς αθώους. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να προβλέψουμε τις ε, ατασταλίες και την, ε, τις καταχρήσεις. Να προωθήσουμε το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, γιατί Θέλουμε οι ζωστοί πληροφο... οι πληροφορίες που θα δίδονται να προστατεύσουν την ε, κοινωνία μας και το κράτος δικαίου και όχι κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει οι προσφεύγοντες να προστατευτούν βάσει των κανόνων του ΟΣΑ, του ΠΟΕ και ούτω καθεξής. περιπτώσει όπως ε, το Panama Papers και άλλες τα τελευταία χρόνια δείχνουν τη σημασία του ρόλου των whistleblowers στην πράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη προστασία τους, αλλά ταυτόχρονα να βεβαιωθούμε ότι οι προσφεύγοντες δεν είναι θύματα αντιπίνων θα πρέπει να αναγνωρίζεται ο ρόλο τους στον αγώνα κατά της διαφθοράς και άλλων, είδου, άλλων είδους ε, εγκλήματα. Οπότε, σε περίπτωση που χάσουν το κύρος τους οι πληροφοριοδότες, να τους δίνουν έντανες εναλλακτικέ. Η κυρία Εστεράς με τις τροπολογίες της έχει τονίσει αυτές τις ιδέες και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να υποβάλει ε, πρόταση για τους πληροφοριοδότες ως το τέλος του χρόνου η πρόταση. Εδώ ίσως αυτό να είναι λίγο βιαστικό. Δεν υπάρχει νομική βάση για να γίνει τέτοια πρόταση. Και έχουμε υποβάλει και άλλη τροπολογία όπου λέμε ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ειδικοί κανόνες για τις πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, άμενα τάξη της διεθνής σχέσης ενός κράτους. Μας αρέσει η ιδέα ενός πολυεπίπεδου συστήματος, ώστε πρώτα να υπάρχει η παράδοση των πληροφοριών εντό ενό οργανισμού ή των αρμόδιων αρχών, ώστε να γίνεται πλήρω σοβαστό το νομικό δικαίωμα και εμπιστευτικότητα και των πληροφοριτών και των ε, ε, δραστών ή όσων έχουν διαπράξει κάτι, ένα δίκημα. Η αντιστροφή του βάρους απόδειξης ε, για να αποδεχθούν τα αντίπεινα από νομικής πλευράς είναι πολύ δύσκολο να το υποστηρίξουμε και να το δικαιολογήσουμε. Δεν μας αρέσει η δυνατότητα ανώνυμης υποβολής εκθέσεων. Είναι σημαντικό να υπάρχει προστασία του απορρίτου, αλλά το να μπορεί κανείς ανώνυμα να καταδίδει μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να προκαλέσει καταχρηστική ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού και γύρει ερωτήματα για το κατά πόσον ε, η αποκάλυψη στοιχείων γίνεται καλόπιστα ή όχι. Και θα γίνεται ε, ολόκληρο θέμα κάθε φορά που υπάρχει η αντίδραση ενός εργοδότη για το κατά πόσον η καταγγελία ήταν καλόπιστη ή θεμητή ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μας μένουν 13 λεπτά για το σύνολο της ε, συνεδρίας σας. Μας μένουν τρία θέματα. Το λέω ως whistleblower, να είστε πολύ σύντομοι. Ευχαριστώ για τις γενικές εισηγήσεις. Ε, συζητήσεις θα ξαναγίνουν και στις 28. Θα έχετε και τις ε, συναντήσεις των σκιωδών ε, στους, ε, στο Στρασβούργο. Ο λόγος στη, στον κύριο Ντυρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ως σκιώδης για τους Πρασίνους. Θέλω από τη μια να θυμίσω όσα είπαμε, αλλά μην ξαναδιαβάσω και όλες τις αρχές που μόλις ακούσαμε και αναγνωρίστηκαν από τις δασικές ομάδες. Απλώς να θίξω μερικά σημεία. Πρώτο, το οποίο θέλω να το πω δημοσίω εδώ και έντονα, ευχαριστώ τη Βρυζινή Ροζιέρ για τη δουλειά που έχει κάνει και τις βελτιώσεις της στις συμβαστικές. Το κείμενο ήταν καλό εξ αρχής, τώρα βελτιώθηκε κι άλλο. Πολύ γρήγορα θα απαντήσω ότι το θέμα της νομικής βάσης είναι πραγματικό, αλλά σε αυτή την ε, φάση στην Ευρώπη βρίσκουμε νομικές βάσεις για το αντίθετο, για να διώξουμε τους ε, whistleblowers που διαρκώς βρίσκονται στα δικαστήρια. Το ανάποδο είναι δύσκολο, να βρούμε βάση για να τους προστατεύσουμε. Εάν θέλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε τους ε, πληροφοριδότες πρέπει να βρούμε νομική βάση. Και να πω με την ίδια ευκαιρία, επειδή η κυρία Φρασόν και ο κύριος Δελτούρα αναφέρθηκαν, ότι τη Δευτέρα μόλις ο Σεμπαστιάν Αρσάκ της LDC 14 ε, διώχθηκε γιατί κατήγγειλε τι σκανδαλώδει ε, συνθήκε εντό των οποίων λειτουργούν κάποιε φαγέ στη Γαλλία. Και γι' αυτό ακριβώ διώχθηκε. Είναι σημαντικό λοιπόν οι πληροφοριδότε να προστατεύονται πολύ γρήγορα για τα σημεία που είναι θέμα για μα. Ε, όχι έρχε. Ο ορισμό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο. Το είπε και εσύ, Βρυζίνη. Πρέπει όλοι οι πληροφοριοδότε να προστατεύονται. Το θέμα τη ανωνυμία. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την ανωνυμία, διότι εξ ορισμού πρέπει να προστατεύουμε ένα πρόσωπο. Εάν ανώνυμη καταγγελία δεν γίνεται κανεί whistleblower εφόσον δεν γνωρίζει κάποια αρχή το όνομά του. Τότε μόνο μπορεί να το προστατεύσει. Οπότε το θέμα τη ανωνυμία νομίζω παραμένει επί ε, τη αρχή θεωρητικό. Επίσης η ιεράρχηση. Εγώ επιμένω από αυτού. Δεν πρέπει να υπάρχει στο σχέδιό μας ιεράρχηση. Διότι ναι, κάποιες φορές μπορεί να πρέπει να κάνει κανείς καταγγελία εσωτερικός, αλλά μερικές φορές δεν γίνεται αν υπάρχει ολοκληρό δίκτυο διαφθοράς. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει ε, η καταγγελία εντός της εταιρεία, θα έπεφτε κατευθείαν ε, η τιμωρία. Πρέπει λοιπόν να μην υπάρξει ιεράρχηση, αλλά να υπάρχει μια αρχή που να λαμβάνει και ανώνυμες ε, προσφυγές, μια αρχή που να ε, λειτουργεί βάσει προποθέσεων. Αυτό ναι, το στηρίζω. Και τελευταία παρατήρηση, το θέμα της καλής πίστης του χρηματισμού. Το δίκαιο δεν έχει καμία σχέση με τις ε, αρχικές προθέσεις των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να κοιτάξουμε τι έχουν στην καρδιά και στο μυαλό τους. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Μπορεί για καλούς ή για κακούς ε, λόγους να κάνουν κάποια κίνηση. Το ερώτημα είναι αν πλήττεται το γενικό συμφέρον. Είναι μια πληροφορία γενικού ενδιαφέροντος. Εάν ναι, ε, είμαστε στην περίπτωση του ε, whistleblower, αν όχι της προσωπικής δυσφήμισης. Ω προ την έννοια τη καλή πίστη, τη γνωρίζουν πολύ καλά οι δημοσιογράφοι. Είναι ένα τρόπο να πούμε ότι ένα πρόσωπο καλόπιστα ζητά ένα θέμα να ληφθεί υπόψη ε, από τις δημόσιες αρχές. Ήμουν στα δυνατόν πιο γρήγορος. Ευχαριστούμε και ο κύριος Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος. Μιλήσαμε για την προστασία των πληροφοριοδοτών και πρέπει να μιλήσουμε επίσης και για τη νομική βάση στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Νομίζω πως πρέπει να απευθυνθούμε στη νομική υπηρεσία και να ζητήσουμε να μας παρουσιάσουν τις επιλογές που έχουμε και να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τη συνεισφορά τους ως τη βάση των συζητήσεών μας. Η ομάδα ECR έχει κάποιες αμφιβολίες για την ε, πρακτική αυτή. Τα κράτη-μέλη καταρχάς πρέπει να, δια... να προστατεύσουν το δικαίωμα των δημοσιογράφων να μην αποκαλύπτουν τις πηγές τους και οι αρχές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους παρακολούθησης για να βρουν τις πηγές. Τώρα, οι καταγγελίες και δεν θα πρέπει να γίνονται για παράνομου σκοπούς ή για να βλάψουν το δημόσιο συμφέρον. Και οι δημόσιε και οι ιδιωτικές επιχειρήσει πρέπει να διαπώνται από συγκεκριμένου κανόνες. Το περιβάλλον πρέπει να έχει κάποιες αξίες. Εάν επιβάλλουμε ορισμένους ε, μηχανισμούς, αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει στην κουλτούρα ορισμένων κράτων μελών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που θα προστατεύουν ε, τους καταγγέλλοντες. Είναι μία σύσταση πιστεύω που η πρόταση μάλλον το να υπάρχει μία ενιαία αρχή είναι υπερβολική. Υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες δεν τηρούν τους κανόνες σχετικά με την προστασία ε, των καταγγελόντων και μάλιστα πολλές φορές ε, ούτε μέσα στην ίδια την Κομισιόν δεν ξέρουν τι ε, γίνεται και ποιοι είναι οι κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άντερσον έχει το λόγο, θα αποσύρω το όνομά μου από τον κατάλογο για ε, χάρη οικονομία χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεμπρετόν έχει το παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προστασία των whistleblowers είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το κοινό συμφέρον. Νομίζω ότι υπάρχει μια συνένεση από αυτού, ε, όπως άλλωστε διαπιστώσαμε και στην χθεσινοβραδινή συνάντηση των σκιών εισηγητών πολλές ε, συμβαστικές προτάσεις θα υποβληθούν. Ε, βεβαίως παραμένουν κάποια ζητήματα. Υπάρχει ένα θέμα νομικής βάσης. Ε, δεν θα πούμε τίποτα από αυτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει την κατάλληλη νομική βάση. Εγώ πάντως ε, θεωρώ ότι η μόνη νομική βάση η οποία ε, αρμόζει ε, η, αυτή του άρθρου 352 της συνθήκης για τις δράσεις, τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης. Βέβαια αυτό τρομάζει πολλούς ε, βουλευτές γιατί χρειάζεται ομοφωνία. Ε, αλλά είναι η μόνη κατά τη γνώμη μου η οποία αρμόζει εδώ. Τώρα, υπάρχει αυτή η ιδέα ότι οι whistleblowers ε, μπορούν να καταγγείλουν όχι μόνο παράνομα αλλά και παράτυπα γεγονότα. Εδώ στο γαλλικό δίκαιο υπάρχει ε, ένας, υπάρχει μια βεβαιότητα, διότι το όρος παράτυπα είναι λίγο προβληματική. Υπάρχει και ο νόμος ΣΑΠΑ 2 στη Γαλλία ε, που μιλάει μόνο για παράνομα ε, γεγονότα, παράνομα, παράνομες πράξεις ε, σε ό,τι αφορά τους και την προστασία τους. τώρα, η καλή πίστη επίσης δημιουργεί πρόβλημα. σε κάποιες χώρες αυτό ενδεχομένως να καταστήσει πιο επισφαλή τη θέση του whistleblower. Ίσως να μπορούσαμε να βρούμε μια άλλη διατύπωση, την οποία όμως θα πρέπει να τη βρούμε. Ε, κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα. Το σκεφτόμαστε. Τώρα το τελευταίο πρόβλημα είναι ότι κατ' εμέ υπάρχουν τρεις τομείς που πρέπει να βρεθούν εκτός του πεδίου εφαρμογής του κειμένου. Ε, το αμυντικό ε, απόρριτο, το ιατρικό απόρριτο και το απόρριτο τον, το δικηγορικό, το δικαστικό, δηλαδή των σχέσεων μεταξύ του δικηγόρου και του πελάτη. Εκεί χρειάζεται, θα χρειαστούν τουλάχιστον είτε εξαίρεση είτε ειδικέ διατάξει. Η Γαλλική Νομοθεσία του 2016 πάντω έχει ε, αποκλείσει αυτού του τομεί. Ε, γενικότερα το κείμενο πάντως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία ε, τονίζονται. Καταρχήν η προστασία δεν θα αφορά μόνο τις εργασιακές σχέσεις. Ε, όχι μόνο αυτοί δηλαδή οι οποίοι είναι εργαζόμενοι κάπου και αυτό είναι καλό διότι στη Γαλλία παραδείγματος χάρη πολύ πρόσφατα η, η γιατρός η Ρεν Φρασόν είχε καταγγείλει τις ε, ε, ε, φαρμάκου χωρίς να διεργάζεται η φαρμακευτική εταιρεία. Ε, δεύτερον, θα υπάρχει ένας μηχανισμός ειδοποίησης σε δύο επίπεδα εσωτερικά στην κάθε επιχείρηση που θα πρέπει να την εθαρρύνουμε να προβλέπει τέτοια διαδικασία και εξωτερικά βέβαια μέσω άμεσης προσφυγής στον τύπο. Βεβαίως, ε, όπως είπε η Πασκάλ Λουρό, ε, μπορεί να επιλέξει ο ίδιος ο whistleblower απευθείας ε, να απευθυνθεί στο ευρύ κοινό, αλλά πρέπει να προβλέπεται και η εσωτερική διαδικασία, διότι πολλοί whistleblowers δεν θέλουν να εκτεθούν στον τύπο. Και αυτή τη δυνατότητα πρέπει να τη δώσουμε. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι η κάθε χώρα θα πρέπει να προβλέψει ε, ένα όργανο προστασία ε, των whistleblowers, ε, όπως θεωρεί αυτή καλύτερα. Πιστεύουμε ότι αυτή η διάταξη σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών. Η προπαρασκευή λοιπόν της έκθεσης ξεκινάει σε καλές βάσεις, χαίρομαι γι' αυτό, θα επαγρυπνούμε για τη συνέχεια σε σχέση και με τις τροπολογίες που έχω υποβάλει. Βεβαίω, εσεί πάντα επαγρυπνείτε, είστε, ειδικεύεστε. Ε, ήθελα κι εγώ να παρέμβω, θα την ακυρώσω όμω όπω και ο κύριο Άντερσον για να μην χάσουμε χρόνο. Ε, η τελευταία συνάντηση άλλωστε πήγε προ αυτή κατεύθυνση, οπότε δεν θα παρέμβω τελικά. Οπότε αν δεν έχετε αντίρρηση, θέλετε ξανά το λόγο. Όχι, πρόεδρε. Ε, η επόμενη συνεδρία του σχεδόν εισαγητών 25 Σεπτεμβρίου και 28 ψηφίζουμε εφόσον όλα πάνε καλά. Μάλιστα, ναι, σίγουρα θα, θα υπάρξουν αιτήματα το 28. Ε, πάμε στο προτελευταίο σημείο της μέσης διάταξης που αφορά την παρέμβαση του κυρίου Αντώνιου Μαριών, Μαριών Πίντο. Παρακαλώ να είστε σύντομος και ο κύριος Λεμπρετό να προλάβει να παρέμβει έγκαιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά να πω για τις τροπολογίες, γιατί ακόμα δεν έχουμε μεταφραστεί. Δεν υπάρχει μετάφραση. Σε κάθε περίπτωση, να ε, εξηγήσω εξ αρχής, ότι ελπίζω να αναβληθεί η ψηφοφορία στη ΛΥΜΠΕ, ώστε να αναβληθεί η ψηφοφορία και στη δική μας Επιτροπή από τις 28 στις 10 Οκτωβρίου. Διότι στις 28 δεν μπορώ να είμαι εδώ. Θα είμαι ε, υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές της Πορτογαλίας στο Δήμο την κοινότητα όπου γεννήθηκα και θα έχω την προεκτική μου εξτατεία. Το πρόβλημα εδώ είναι το εξής. Δεν θεωρώ ότι είναι δυνατό να υλοποιήσουμε ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χωρίς πραγματική ολοκλήρωση στο χώρο τη δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, ομοιόμορφη. Δεν λέω ομογενή. όλες οι υποθέσεις να εκδικάζονται με τον ίδιο τρόπο στις χώρες, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας βασικός πυρήνα αντικειμάτων, ο οποίο να έχει την ίδια μεταχείριση σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, υποθέσεις που τις χειρίζονται τελείως διαφορετικά οι χώρες μεταξύ τους, αυτό δεν μπορεί να γίνεται πλέον. Και επίσης υπάρχει και ε, οργανωμένη εγκληματικότητα σε επίπεδο εμπορίου όπλων, ανθρώπων, ναρκωτικών, οικονομικού εγκλήματος, φόρα αποφυγής, ε, διαφθοράς, λεύκανσης, παράνομων προσόδων. Αυτά είναι εγκλήματα ενωσιακού ε, βεληνικούς και πρέπει να τα βλέπουν όλα τα κράτη με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον χώρο της δικαιοσύνης. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εισαγγελία. Και το Ευρωκοινοβούλιο να έχει ένα σημαντικό ρόλο εδώ να διαδραματίσει, ένα ρόλο ε, κεντρικό στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι αποτελεσματική, ότι λειτουργεί εύρυθμα, ότι είναι ανεξάρτητη. Να μην είναι απλώς ένα πολιτικό εργαλείο που να το χειραγωγούν οι πολιτικοί ηθήνοντες ή τα κράτη-μέλη. θα πρέπει και για την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κοιτάξουμε να μην ισχύσουν οι παρόμοιοι κανόνες με τα δικαστήρια ορισμένων κρατών μελών όπου διορίζονται δικαστές και μοιάζει να έχουν γίνει κολέγιο των επιτρόπων. Ε, θα πρέπει λοιπόν και στην Ευρώπη να κοιτάξουμε να δημιουργηθεί μια εισαγγελία η οποία να είναι πραγματικά εισαγγελία δικαιοσύνης με ανθρώπους που να προωθούν τη δικαιοσύνη και όχι απλώς να κατηγορούν ε, σύμπαντες όλους με κάθε τίμημα, θα πρέπει να προωθείτε η δικαιοσύνη, να πηγαίνουν στα δικαστήρια υποθέσεις που αξίζει να, εκδικαστούν και να λαμβάνουν μια ανεξάρτητη μερόληπτη απόφαση οι δικαστές. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσει και να υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είχα πάρα πολλά να πω, αλλά το πλέον σημαντικό νομίζω ήταν αυτό. Το Ευρωκοινοβούλιο, αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να έχει ένα σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της εισαγγελία και κυρίως στην εξασφάλιση της ανεξάρτητης λειτουργίας της εισαγγελία ώστε να μην είναι ένα πολιτικό εργαλείο στα χέρια των ε, πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών. Ευχαριστούμε πολύ και για την ουσία και για την ταχύτητα τη παρέμβαση. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνιο. Ο κύριος Φως, γρήγορα παρακαλώ και εσεί. Ναι, γνωρίζω πόσο λίγο χρόνο διαθέτουμε. Θα ήθελα όμως να τονίσω δύο σημεία. Καταρχάς να πω ότι στηρίζω την συγγήτρια γιατί πρέπει όντω ε, να ε, ξεκαθαρίσουμε ποιες αρμοδιότητες θα έχει η Eurojust και ποιες η ΕΠΟ. Και μετά σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, νομίζω πως εδώ θέλει προσοχή διότι χρειάζεται προσαρμογή των ε, διατάξεων σχετικά με την προστασία δεδομένων σε αυτά που έχουμε μέχρι τώρα ε, καταφέρει. Ίσως ε, αυτό είναι και το σημαντικότερο επίσης, να δούμε δηλαδή αν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ε, και με το Διοικητικό Συμβούλιο και με, το, ε, με τους άλλους ε, αρμόδιους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και από μένα και από τους διερμηνείς ευγνωμοσύνη μας. Το θέμα το εξαντλήσαμε. Θέλει και άλλο το λόγο, κύριο ναι, ευχαριστώ Ζαμαρή πολύ πολύ γρήγορα για να πω ότι στρίζουμε πολύ την τοποθέτηση του κυρίου Πίντο ε, και την τάση της έκθεσης και μας ενδιαφέρει πολύ η ανεξαρτησία ε, και η μη ε, δημιουργία σχέσεις μεταξύ Eurojust και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. να πω λοιπόν ότι στηρίζω την εξαιρετική έκθεση του κυρίου ε, Μαρνιού κυρία Κάουφμαν παρακαλώ πολύ γρήγορα. Äh, και εγώ Θέλω να ευχαριστώ τον εισηγητή, του και εισηγητές εκ μέρους της δική μας ομάδας να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Eurojust να προσαρμοστεί στο γενικότερο κόνσεπτ των ευρωπαϊκών οργανισμών. Είναι σαφές πως είναι πολύ σημαντικό οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Eurojust να είναι συμβατές μεταξύ τους και φυσικά χρειάζεται να δούμε το θέμα του κεντρικού ε, συντονισμού, να δούμε και τον τρόπο εργασίας των ε, οργανισμών. Γι' αυτό λοιπόν ε, χαίρομαι των προτέρων για την ε, συνεργασία με τον εισηγητή και τους Σκιώδης. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Να δούμε τώρα το χρονοδιάγραμμα, ακόμη και αν είναι λίγο πιεστικό, θα πρέπει το σεβαστούμε. Το τελευταίο σημείο 22 μας το παρουσιάζει ο κ. Λεμπρετό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για εκτελεστικές πράξεις, κλασικές εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής για την ε, τήρηση των, Ευρωπαϊ... διεθνών λογιστικών προτύπων. Θα πρέπει να τα σεβαστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρμόδια καθ' η, Ευρωπαϊκή... η Επιτροπή ε, οικονομικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 106 πρέπει και εμείς να βεβαιωθούμε ότι ε, δεν αντίκειται τίποτα στο δίκαιο της Ένωσης από τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχω τίποτα να παρατηρήσω επί του κειμένου, δεν υπάρχει παρέμβαση των αρμοδιότητων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κάτι που να αντιφάσχει με το ενωσιακό δίκαιο. Και ξέρουμε ότι και σε αυτό το τομέα είστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικός. Είμαι ιδιαίτερα προσεκτικό κύριε Πρόεδρος και ε, θα σα επισημάνω, μια και με αφήσατε, ότι αν είχατε αφήσει περισσότερο χρόνο θα έλεγα και για την περισσότερη προηγούμενη έκθεση κάτι, αλλά κοιτάξτε να μην σύντομο. Ναι, να δώσω τρει ε, πληροφορίε τώρα. 28 Σεπτεμβρίου 2017, επόμενη συνεδρίαση. Ε, πραγματικά ρηξικέλευτη είδηση. Επίση, να ευχαριστήσω του διερμηνεί, οι οποίοι μα έδωσαν κάποια περιπέτεια λεπτά. Και τρίτον, θα έπρεπε να ξεκινήσω αυτή τη συνεδρία ρωτώντα αν περάσατε καλά τι διακοπέ σα, κάτι που ήταν ε, προφανέ, διότι σεβαστήκαμε πλήρω τον χρόνο τη συζήτησή μα ε, και τα καταφέραμε. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Μπερζερόν που μετέφερε τα λόγια μου. Ε, καλή σα ημέρα. Αυτό το απόγευμα δεν θα υπάρξει συνεδρίαση.